Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Uh, Δεν χρειάζεται να σας κάνω συστάσεις. Να πω παρόλα αυτά ότι είναι εδώ ο Φρανς Τίμερμανς, που είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος ε, στη νέο εκλεγήσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιοι από εσά συμμετείχατε και στις ε, ακροάσεις, επομένω δεν είναι και η πρώτη φορά που γνωρίζεστε με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν. Ε, εχθές ε, συνεδρίασε ουσιαστικά η πρώτη ε, για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε όμως, επειδή ακριβώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε όλα όσα θέλουμε ε, στη διάρκεια των ακροάσεων, να κάνουμε μια σύντομη συνάντηση, να μας πείτε δύο λόγια για το πώς βλέπετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πρώτες μέρες και ε, να μας πείτε και πώς βλέπετε λίγο το μέλλον. Ε, επίσης, ε, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα θέματα τα οποία είναι τμήμα της αρμοδιότητας της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων βεβαίως, αλλά οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, πρόσδεκτο. Θα δώσουμε λοιπόν τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς και μετά πάρα πολύ πειθαρχημένα, γιατί έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ, προκειμένου να κάνουμε διάλογο. Δεν είναι ακρόαση, το λέω συνέχεια στον εαυτό μου αυτό, διότι ε, έχω πρόσφατη εμπειρία ακρόασης, αλλά είμαι εδώ για να τίνω ευήκο σε αυτά που έχετε να πείτε εσείς, να μου πείτε τις ιδέες σας για το πώς θα συνεργαστούμε τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι ε, εγώ και εσείς θα συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά για διάφορους λόγους, αλλά θα ήθελα εν συντομία να σταθώ στο πιο σημαντικό θέμα, το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το προετοιμάσω αυτό πολύ σύντομα και θα προτείνω και σχετική συζήτηση από αυτού και στο Σώμα των Επιτρόπων και στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να βεβαιωθώ ότι το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αντανακλά σαφέστατα τη συμφωνία που έχει κάνει ο πρόεδρος Γιούνκερ με το κοινοβούλιο σας στις 10 βασικές προτεραιότητες. Και θέλω το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντικατοπτρίζει σαφέστατα αυτές τις 10 προτεραιότητες και θέλω ο κάθε επίτροπος όταν θα προετοιμάσει τη συνεισφορά του στο πρόγραμμα εργασίας να επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε αυτές τις 10 προτεραιότητες. Διότι αν θέλουμε να αλλάξει ο τρόπος εργασίας, γιατί αυτό θέλουμε και να κάνουμε, διότι είδαμε και τι είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ από αυτού, είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει τα πράγματα και να κάνει διαφορετικά πράγματα. Και αυτό θέλουμε να αντανακλάται ήδη στο πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη χρονιά. Και φυσικά εκεί θα επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες που καθορίσαμε και συμφωνήσαμε με το Κοινοβούλιο. Και με βάση αυτές ε, ε, υπερψηφίσατε κι εσείς αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό ακριβώς ε, καθήκον μου είναι να βεβαιωθώ ότι η ψήφος αυτή και η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε για να υπάρξει αυτή η ψήφος ε, θα υλοποιηθεί. Δεν θα επικεντρωθούμε μόνο σε αυτές τις 10 προτεραιότητες, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και ε, λίγο πώς να εργαστούμε με διαφορετικό τρόπο ε, ξέρετε ότι το θέμα των αντιπροέδρων και οι επιπλέον αρμοδιότητες έχει δημιουργήσει ερωτηματικά στο Κοινοβούλιο και τώρα καθήκον έχουμε να σας δείξουμε ότι θα λειτουργήσουμε καλύτερα από ό,τι οι προηγούμενες επιτροπές. Αυτό βέβαια θα φανεί στην πράξη αυτό που είδα εγώ στη διάρκεια της πρώτης μου εβδομάδας και κατά την προεσημασία για αυτή την πρώτη εβδομάδα είναι ότι όλοι οι επίτροποι ε, είναι καθόλου διατεθειμένοι να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό το σύστημα διότι μόνο έτσι η προτεραιότητα θα μπορέσει να θέσει προτεραιότητες, να επικεντρωθεί στις προτεραιότητες και αν μου επιτρέπετε να είναι και λίγο πιο πολιτική από ό,τι στο παρελθόν υπό την έννοια ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γεννήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν αυτό δεν θα πρέπει να διαφαίνεται μόνο στο πρόγραμμά μας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε από τούδε και στο εξή. Και εδώ έρχομαι και σε κάτι άλλο, παρόλο που γνωρίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν και να ολοκληρωθούν, αλλά αυτό θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα προετοιμάζουμε το έργο μας και το πώς θα προετοιμάζουμε την νομοθεσία και υπάρχει μια προνομική σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτήν θα την ε, θεμελιώσουμε περαιτέρω, αλλά ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, συμπεριληφθεί και το Συμβούλιο στην ε, διαδικασία προετοιμασίας και εκτέλεσης του προγράμματος και στον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε. Διότι αυτό διαφαίνεται και από τη συνθήκη. Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών εργάνων κατά την εκτέλεση όσων έχουν συμφωνηθεί από εμάς σε πολιτικό επίπεδο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τη θέση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ θεωρώ και για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Συμβούλιο, δεν αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γιατί αυτό είναι διαφορετικό θέμα, το Συμβούλιο να συμμετέχει περισσότερο στην προετοιμασία και την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας ε, της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό εν είδη σύντομης εισαγωγής, ε, σας είπα ότι θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και επειδή ακριβώς θέλω να έχουμε διάλογο και δεν θέλω να κάνουμε πάλι ακρόαση, να δώσω και πάλι τα ενία στην Πρόεδρο. Συνάδελφοι, Έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας για τις συζητήσεις. Ζητήσαμε από τους συντονιστές σας να σας ενημερώσουν ότι μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις, όχι όμως για πάνω από τρία λεπτά. Και ο Σέπλιν για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω, κύριε Αντιπρόεδρε. Είναι τιμή μας γιατί είμαστε η πρώτη επιτροπή την οποία επισκέπτεστε και θα ήθελα να θέσω ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες ε, συνεχίζουν την εισαγωγή την οποία κάνατε με πολιτικό τρόπο. Καταρχάς η πρώτη ερώτηση, η πρωτοβουλία των πολιτών. Ξέρετε ότι πέρασε από μας ε, η μέθοδος αυτή και ανησυχούμε για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Και διορθώστε με, υπήρξαν 17 τέτοιες πρωτοβουλίες, μόνο μία έχει γίνει δεκτή από δημοσκοπήσεις τις οποίες κάναμε, οι κανόνες είναι πάρα πολύ αυστηροί και πολύ περιοριστικοί και ερμηνεύονται ακόμα και πιο περιοριστικά. Η ερμηνεία που δίδεται είναι περιοριστική και δεσμευτική. Εγώ δεν λέω ότι ε, είναι εύκολο πράγμα. Προφανώς σε οργανωτικό επίπεδο είναι δύσκολο ε, να συλλέξει κανείς ένα εκατομμύριο υπογραφές. Αλλά η απόρριψη μιας τέτοιας διαδικασίας ε, δυστυχώς ρίχνει, λάδι στη φωτιά του αντιευρωπαϊσμού. Νομίζω ότι πρέπει να μας δώσετε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει η πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο να πιστεύει ότι είναι άχρηστη η δυνατότητα, η πιθανότητα επηρεασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η New York Times χθε, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, ε, είχε κύριο άρθρο ε, από την αρχή συνταξία, ασκώντας κριτική άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Jean-Claude Juncker, ο πρόεδρος της Επιτροπής, θα πρέπει να ασκήσει την αρμοδιότητά του και να υποχρεώσει τον κύριο Ναύρασιτς να παραιτηθεί. Αυτό είναι ένα άρθρο εφημερίδας, εντάξει. Βέβαια από μια εφημερίδα πολύ σημαντική, όχι άμεσα εμπλεκόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, αλλά παρόλα αυτά είναι μια άμεση ε, εμπλοκή ε, στις διαδικασίες ε, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε ψηφίσει για το συγκεκριμένο πρόσωπο και παρεμβαίνουν ε, με έμεσο τρόπο λέγοντας ότι οι Ούγγροι δεν πρέπει να έχουν επίτροπο. Δεν ξέρω τι σχόλιο μπορείτε να κάνετε σε αυτό. Και τρίτο, γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ανεπίσημη ομάδα βουλευτών που ασχολείται με την ε, συμφιλίωση των ευρωπαϊκών ιστοριών. Συναντηθήκαμε χτες και βασική μας ε, ανησυχία είναι η αποκατάσταση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στα προηγουμένως κομμουνιστικά κράτη. Αυτό έχει σχέση και με τα εγκλήματα του κομμουνισμού που πρέπει να ερευνηθούν αυστηρά και το ίδιο αφορά επίσης και τα εγκλήματα του ναζισμού. Είναι κάποια από αυτά εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας και αν και πρέπει να επιμείνει κανείς ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το καθολικό, τότε θα πρέπει να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας θυμίσω συνάδελφοι ότι θα πρέπει να παραμείνετε μέσα στο τρίλεπτο μπρέσο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη για να μπορέσει και άλλο μέλος της ομάδας μου να πάρει το λόγο. Θα ομιλήσω την Ιταλική την οποία κατέχετε. Better regulation, καλύτερη νομοθετική δραστηριότητα. Ε, ξέρετε, εσείς αναφερθήκατε πολύ γενικά σε αυτό στην εισαγωγή σας θα ήθελα να μου πείτε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να εργαστείτε. Ε, καλύτερα σημαίνει και λιγότερο, θέλετε κάτι να απλωστεύσετε μόνον ή κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει πώς ακριβώς πιστεύετε ότι θα πρέπει επίσης να συνεργαστείτε και με την Επιτροπή μας. Το δεύτερο θέμα, ίσως αν είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε και μια άλλη φορά, ε, μου έχετε πει, κατά τη διάρκεια της ακρόασης εννοώ, ότι θα πρέπει να προσπαθήσει κανείς να εργαστεί έτσι ώστε να εφαρμοστεί όσο περισσότερο γίνεται η συνθήκη της Λισαβόνας πριν αρχίσει κανείς να σκέφτεται διαφορετικές αλλαγές, βελτιώσεις κτλ. Λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς και σε ποιους τομείς και σε ποιους χώρους βλέπετε ότι υπάρχει χώρος για καλύτερη και περισσότερη εφαρμογή γιατί εμείς ε, προετοιμάζουμε μια έκθεση για τη συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύετε ότι εδώ είναι θέμα προσωπικό, πιστεύετε δηλαδή ότι θα πρέπει να ερευνήσουμε σε βάθος και την αρχή της επικουρικότητας, έτσι ώστε να, αν όχι καταργηθούν, εν πάση περιπτώσει να μικρύνουν κάποιες περίπλοκες ρυθμίσεις νομοθετικές. Σας ευχαριστώ και τώρα να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονικό όριο των τριών λεπτών. Για το ECR τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να μιλήσω πολυνικά. Grupie Στην ε, ομάδα μας, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι οι νομοθεσίες ε, των εθνικών κοινοβουλίων και τα δικαιώματα των πολιτών. Ω εκ τούτου, λοιπόν, να σα ε, θέσω τα ερωτήματα που έχω να σα κάνω. Είσαστε αντιπρόεδρο πλέον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε εκφράσει ιδέε και σαφέστατε απόψει και τοποθετήσει για τι νομικέ πράξει και για το ποιε εξ αυτών θα έπρεπε να αποσυρθούν. Για παράδειγμα, για να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας. Και για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από υπερβολικά μεγάλη κεντρική διαμόρφωση των πολιτικών. Ποιες λοιπόν θα ήταν αυτές οι νομοθετικές πράξεις. Οι νομοθετικές πράξεις που θα έπρεπε να καταργηθούν για να μην υπάρξει παράβαση της επικουρικότητας. Ήθελα επίση να σα ρωτήσω το εξή Σε ό,τι αφορά την πολιτική σας δράση, τι θα γίνει αν κάποια εθνικά κοινοβούλια ταχθούν ηχηρά κατά κάποιας νομοθετικής πράξης γιατί θεωρούν ότι αυτή παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Ποια θα ήταν η δική σας αντίδραση στην περίπτωση αυτή. Θα αντιδρούσατε με πολιτικό τρόπο ή θα επικαλεστείτε τη δυναμική βάση. Και αυτό με οδηγεί και στην επόμενη ερώτησή μου. Την οποία ήδη και ακούσαμε ένα θέμα που έθεσε συνάδελφος. Είπατε εσείς ο ίδιος ότι ακόμα και αν αναπευθεί η πρωτοβουλία των πολιτών δεν θα έχει τερματιστεί ο Βρετανικός διάλογος. Πώς θα διαμορφωθεί λοιπόν ο διάλογος αυτός σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή η οποία έλαβε ευρεία υποστήριξη. Πώς θα διαμορφωθεί λοιπόν συγκεκριμένα αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Sí, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τίμερμανς, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Εσείς ε, έχετε διευκρινίσει σε αρκετές περιπτώσεις ότι είστε αποφασισμένοι η συνθήκη της Λισαβόνας να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν εν μέρη αλλαγές και ποιοι τομείς είναι αυτοί οι οποίοι θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να εξετάσετε και θα μπορούσατε να τροποποιήσετε μερικώς. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της εξωτερικής εκπροσώπησης της Ευρωζώνης. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ξέρουμε ότι δημιουργεί σε κάποιες χώρες περισσότερους δισταγμούς από όλους. Ζητούν να αυξηθεί αυτή η ευρωπαϊκή φωνή και θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον είχατε ε, ήδη τη δυνατότητα να σκεφτείτε με ποια μέσα θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτούς τους δισταγμούς και να αυξήσουμε την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης. Και τρίτον, θα ήθελα να δούμε αν μπορούμε να είμαστε πρακτικοί σε ένα θέμα το οποίο είναι όλο ένα και πιο σημαντικό. Ο κύριος Μπούτρος Γκάλι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, το 1992 επεσήμανε ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι ε, θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον έλεγε τότε ότι εάν κάθε μία από τις εθνοτικές, θρησκευτικέ ή γλωσσικές ομάδες ε, είχε ε, προσδοκίες για καθεστώς κράτους, δεν θα υπήρχε ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική πρόοδος, θα ήταν όλο ένα και πιο δύσκολο να τη διασφαλίσουμε. Αυτή τη στιγμή, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένες φορές υπάρχουν ε, ανεπίσημες ή και ανεύθυνες θέσεις για το ενδεχόμενο ε, πιθανής απόσχησης συγκεκριμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και αντί να ε, ε, ασχολούμαστε με τα σημαντικά θεμελιώδη ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται αυτό το ζήτημα το οποίο αφορά και το τι αποτελεί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια θέματα θα μπορούσαν να είναι πιο σημαντικό. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε πιο δραστήριοι και θα ήθελα να ακούσω και τι άποψη έχετε εσείς από αυτό. Ο κύριο Κατρούγκαλο εκ μέρου Ενωτικής Αριστεράς. Have... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και τη σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια σειρά αποφάσεων τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων που εποπτεύει τον κοινωνικό χάρτη που έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι παραβιάζει η Ελλάδα τον κοινωνικό χάρτη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος ε, λιτότητας που προβλέπουν τα μνημόνια. Είχαμε επίσης μια έκθεση του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης που επίσης υπογράμμισε ότι πολλές πτυχές της πολιτικές αυτές είναι επιπαραβάση βασικών θεμελιωδών αρχών και επιπλέον είχαμε και δύο εκθέσεις, μία γενική και μία πιο ειδική για την Ελλάδα του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών που επίσης ε, τόνισε ότι οι πολιτικές λιτότητας των μνημονίων παραβιάζουν πολλές συνθήκες του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων και το σύμφωνο για τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσπάθησε να μην απαντήσει άμεσα τα ερωτήματα αυτά, δηλώνοντας ότι οι πολιτικές λιτότητας των ε, μνημονίων δεν αποτελούν δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επιτρόπος Κατάινεν επίσης απάντησε σε σχετική ερώτηση την οποία του απέφθηνα ότι για τον λόγο αυτό ούτε ο θεμελιώδης χάρτης ε, των ανθρωπινών δικαιωμάτων της συνθήκης Λισαβόνας ισχύει. Πιστεύετε σοβαρά ότι σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αυτές και υπό την επιτήρηση δύο θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μπορεί κανείς να διατείνεται ότι δεν ισχύει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σοβαρό να λέμε ότι για κάποιες χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό τα προγράμματα αυτά δεν ισχύει ο χάρτης των ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και να σχολιάσω επίσης το θέμα της αιρεσιμότητας που συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα αυτά σε τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα, όπως για παράδειγμα το εργασιακό δίκαιο. Όπως τα ξέρετε κατά πάσα πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ε, πιέζει την ελληνική κυβέρνηση να νομιμοποιήσει εκ νέου πράγματα τα οποία δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα. Τις απεργίες εργοδοσίας. Εκεί δεν υπάρχει πολιτική από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να επιβάλλεται μια τέτοια πολιτική ατζέντα νεοφιλελεύθερη πασιφανώς σε μια χώρα της Ένωσης. Και το ερώτημά μου, το πιο ουσιώδες, είναι πώς θα αλλάξει η κατάσταση, πώς σκοπεύετε να αλλάξετε την κατάσταση, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν συνδέονται με τους κανόνες διακυβέρνησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci, Madame la Ευχαριστώ, Πρόεδρε. είχατε κάνει την τιμή να μου απαντήσετε γαλλικά στην ακρόαση και θα το κάνετε πάλι, είμαι βέβαιος. Θα είμαι λίγο μονότονος ή μονοθεματικός καλύτερα, έχω θέσει το ερώτημα ήδη, αλλά είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία έχετε συζητήσει και ο κύριος Γιούνκερ, είναι το θέμα της διαφάνειας. Της διαφάνειας στα πλαίσια της λειτουργίας σας. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε λέγοντας ότι η διαφάνεια είναι ένα από τα κλειδιά, δεν είναι η λύση, αλλά είναι ένα από τα κλειδιά της συμφιλίωσης των Ευρωπαίων πολιτών με τα ευρωπαϊκά όργανα. Η διαφάνεια λοιπόν είναι μια προϋπόθεση λειτουργίας της δημοκρατίας, δεν είναι μια επιλογή. Οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι γενικότερες ε, ε, προβληματικές για τη λειτουργία των οργάνων. Δεν θα τα συζητήσουμε όλα τώρα, αλλά υπάρχουν κάποια επιμέρους σημεία τα οποία παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον. Στην χάρτα των επιτρόπων υπάρχει το θέμα των προσωπικών συμφερόντων και των οικογενειακών συμφερόντων. Υπάρχει μια διχοτομία. Στη δήλωση υπάρχει η λεγόμενη προσωπική δήλωση συμφερόντων ενώ αντίθετα στη χάρτα μας λέγεται ότι θα πρέπει επίσης να μην ασχολείστε με θέματα όταν υπάρχουν οικογενειακά συμφέροντα οικονομικά. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια διευκρίνηση που πρέπει να γίνει, εσείς σαν πρώτος αντιπρόεδρος. Ξέρετε θα απαντήσετε, αλλά θέλω να τα ακούσω να το λέτε. Ε, ότι δεν θα υπάρξει ε, κάποια δυσκολία σε σχέση με τα οικογενειακά συμφέροντα. Δεύτερη ερώτηση. Θα συμφωνήσετε μαζί μου λέγοντας ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ε, συνέπεια που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που λέει η χάρτα των επιτρόπων και στις αρχικές δηλώσεις. Η δεύτερη ερώτηση τώρα είναι πολύ πιο σύντομη. Είναι ο κατάλογος στο Μητρό των Λόμπι. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό πάρα πολλές φορές Ξέρετε ότι είναι υποχρεωτικό ε, και για τον Επιτροπή και για το, είναι, για το Κοινοβούλιο. Ε, το Συμβούλιο τι γίνεται. Είχαμε μιλήσει για μητρό διοργανικό, το είχε συζητήσει ο κύριος Γιούνκερ. Μπορεί να κάνω και λάθος, διορθώστε με, είμαι νέος εδώ. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Συμβούλιο αν χρειαστεί να περάσουμε και από μια νομοθετική διαδικασία. Δεν ξέρω αν συμμερίζετε τους φόβους μου. Αντινόλφη για τους φιλελευθέρους. Για την διαφάνεια, εμείς με την ομάδα μας καταθέσαμε ορισμένες τροπολογίες έτσι ώστε να καταστήσουμε υποχρεωτική με ονομαστική ψηφοφορία την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής και να ακυρώσουμε τους κανόνες που προβλέπουν μυστικές ψηφοφορίες για την επικύρωση των επιλεγμένων επιτρόπων για να υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στις δηλώσεις από τη μία τις γενικές, τις δηλώσεις επί της αρχής και τις συγκεκριμένες ενέργειες από την άλλη. Αυτά αφορούν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και τη λειτουργία των οργάνων μας. Θα μιλήσω Ολλανδικά μαζί σας γιατί δεν είναι τόσο καλά τα Ιταλικά μου. Ερώτω πώς αντιμετωπίζετε τη νέα κατάσταση γιατί αντίθετα με παλιότερα που ήμασταν προσανατολισμένοι μεταξύ ΕΛΚ και Σοσιαλιστών και αυτό αποτυπωνόταν και στις προεδρίες του Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή, πλέον υπάρχει μια νέα ισορροπία. Εσείς ως δημοκράτης ε, θα πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη μεταξύ ε, φεντεραλιστών και συμφεραντιλιστών. Εδώ στο Κοινοβούλιο οι συμφεραντιλιστές όπως και εγώ όπου θέτουν ε, την έμφαση στο Συμβούλιο, στα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο που θα πρέπει να δράσει κτλ. Όλα αυτά είναι καινούργια εδώ. Και από την άλλη έχουμε τους φεντεραλιστές ε, οι οποίες ε, μιλούν και αποφασίζουν. Η δημοκρατία ε, και εσείς ανήκετε σε αυτό το δημοκρατικό σύστημα. Πατάτε πετάλι για να προχωρήσει η δημοκρατία στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αν συνεχίσουν τα πράγματα όσα έχουν σήμερα, μετά βλέπουμε ότι όλο και πιο πολύ αυξάνονται οι τομείς της πολιτικής, οι τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς τα επιτρέπετε όλα αυτά. Το ερώτημα λοιπόν είναι... Η δημοκρατία είναι 50 συν 1, αλλά και το να ακούμε νέε τάσει. Εσεί σε τι βαθμό είσαστε πρόθυμο να ακούσετε αυτέ τι νέε τάσει και να σηκώσετε το πόδι από το γκάζι και να σκεφτείτε τις ε, αρμοδιότητες της καινούργιας, τους καινούργιους τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ακούσαμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Να δούμε πόσο χρόνο θα έχουμε και για το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Εξαρτάται πόση ώρα θα μου πάρει. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει αν μπορώ και θα σας δώσω μια ειλικρινή απάντηση αν μπορώ, είτε γιατί δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα ή γιατί πρέπει να το συζητήσουμε εσωτερικώς. Ε, είμαστε στις αρχές ακόμα, τέταρτη μέρα της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, δύο ερωτήσεις. Είχαμε γι' αυτό και ο κύριος Βογιαστόφσκι ήταν σαφέστατος. Ε, αναφέρθηκε σε αυτό που είπα στη διάρκεια της ακρόασης. Και πιστεύω ακράδαντα ότι ήμασταν πολύ τυπολάτρες εδώ. Υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία και αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις τότε η νομική απάντηση είναι απάλλητα σαφής, δεν μπορεί να προχωρήσει η πρωτοβουλία. Όμως, θα μπορούσα ίσως να προβλέψω μια περίπτωση στην οποία ακόμα κι αν δεν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για να προχωρήσει η πρωτοβουλία των πολιτών, το γεγονός ότι τόσοι πολίτες μπήκαν στον κόπο να εκφράσουν την άποψή τους, να υπογράψουν ένα έγγραφο και θέλουν η Ευρώπη να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, θα πρέπει να αποτελεί από επαρκέ κίνητρο για αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ξεκινήσει τουλάχιστον ένα πολιτικό διάλογο επί του ζητήματο. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι εσείς ως εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού λαού θα πρέπει να συμμετέχετε αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία και θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον τη δυνατότητα να κάνετε ένα πολιτικό διάλογο επί του ζητήματος υπό τη μορφή ακρόασης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. Τα εξέτασα όλα αυτά κατά την προετοιμασία για την ακρόαση και δεν βρήκα ε, πουθενά λάθος σε οποιαδήποτε απόφαση έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, κανένα λάθος από νομική σκοπιάς, αλλά είχα συνεχώς την αίσθηση ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε την πολιτική ευκαιρία να κινητοποιηθούν οι πολίτες και να πούν στην Ευρώπη «Ε, «Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μας ικανοποιεί, θέλουμε να το συζητήσουμε». Την ευκαιρία δηλαδή να συμμετέχει κάποιο ενεργά σε μια συζήτηση με το τμήμα τη Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης που ενδιαφέρεται για το ζήτημα αυτό. Ε, έτσι θα το παρουσιάσω στους συναδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα αλλάξω και να σας πω ότι δεν θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Οι κανόνες είναι κανόνες και εμείς είμαστε θεματοφύλακες της συνθήκης και των κανόνων. Δεν μπορούμε να τους παρακάμψουμε. Επομένως, ίσως η πρωτοβουλία αυτή δεν μπορεί να υποστηριχθεί βάσει κανόνων, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσει ένας πολιτικός διάλογος για κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους. Δεν είδα το άρθρο στους New York Times ε, για τον ε, συνάδελφό μου, τον Επίτροπο Ναυράτσιτς, να σας πω το εξής όμως. Δεν αποφασίζουν οι New York Times για το ποιο θα είναι επίτροπο και ποιοι θα είναι επίτροποι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει. Και εσεί ψηφίσατε ε, τη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για τα κράτη-μέλη, θα απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένα σε αυτές τις ερωτήσεις. Στις αρχές της εβδομάδας συναντήθηκα με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας και του το είπα. Εάν προκύψουν ζητήματα, τότε θα εξετάσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα και θα ε, γίνει διάλογος επ' αυτού και θα είμαστε πάρα πολύ ακριβείς. Και αυτός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και το αυτό ισχύει και για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλα τα κράτη-μέλη και για τα 28. Όλοι έχουν το δικαίωμα να προσεγγίζονται τα ζητήματα με τον ίδιο τρόπο. Αν υπάρχει πρόβλημα και δεν επιλύεται, λαμβάνονται μέτρα τα οποία έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει διαδικασία επιπαραβάση ή κατάσταση. Αλλά χωρίς προκατάληψη και με πολύ ακριβή νομικό τρόπο. Εάν ε, οι υπόλοιποι θέλουν να κάνουν μία ε, έντονη πολιτική συζήτηση επί του ζητήματος, υπάρχουν άλλα βήματα στα οποία μπορούν να γίνουν αυτά. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι ακριβής, ε, πρέπει να βασίζεται στους νομικούς κανόνες, στις συνθήκες και στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι ο καθένας είναι υπόλογος ενώπιον αυτών των υποχρεώσεων. Όσον αφορά την συμφιλίωση της ευρωπαϊκής ιστορίας, ε, και πάλι αυτό το ζήτημα είναι πολιτικής φύσεως. Αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική και για μένα από προσωπική σκοπιά. Θυμάμαι ακριβώ πριν από 25 χρόνια ότι δεν μπορούσα να μείνω στι κάτω χώρε. Ήθελα να πάω στο Βερολίνο να δω τι γίνεται εκεί. Και προσπαθώ να το πω και στα παιδιά μου που δεν το έχουν βιώσει αυτό. Ο μεγαλύτερο γιο μου γεννήθηκε το 1989. Ότι άνθρωποι που τους βλέπετε τώρα και είναι στην αίθουσα και είναι Ευρωπαίοι όπως όλοι εμείς, μέχρι τότε ζούσαν σε μια καταπιστική κοινωνία που δεν τους επέτρεπε να εκφράζουν την άποψή τους, τους φυλάκιζε όταν εξέφραζαν την άποψή τους και θεωρώ ότι ο καθής από εμά θα πρέπει ε, να αφιερώσει δύο ώρες να δει τις ζωές των άλλων για να καταλάβει πώς ακριβώς ήταν η καταπίεση σε αυτή την κοινωνία που ζούσε αυτή την ε, ε Εγώ δεν έχω καμία νοσταλγία για την Ανατολική Γερμανία και νομίζω ότι κανένας δεν θα έπρεπε να έχει νοσταλγία για την Ανατολική Γερμανία. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στη ζωή μου που να θα είναι ποτέ πιο σημαντικό από αυτό το ε, χάσμα των δύο Ευρώπη, οι δύο Ευρώπες οι οποίες χωρίστηκαν ακριβώς από την ιστορία. Και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας για να αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι στην ανθρώπινη φύση που προσκαλεί τη δικτατορία όταν δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί και όταν δεν εφαρμόζουμε πλήρως το κράτος δικαίου. Και αυτό με οδηγεί σε μια άλλη ερώτηση για το κράτος δικαίου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε κράτος μέλος να είναι υπόλογο για κάθε εξέλιξη στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Κάθε κράτος μέλος ε, υπέγραψε και κύρωσε τη χάρτα των θεμελιωδικών δικαιωμάτων. Έχει ε, υπογράψει και έχει επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ήγηκε η ώρα να συμμετέχουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να είναι υπόλογο να εφαρμόζει τους κανόνες της χάρτας και της σύμβασης. Και θεωρώ και η πολύ συγκεκριμένη ερώτηση ε, που ετέθη για την Ελλάδα, να έρθω και σε αυτήν, η Ελλάδα ως κράτος μέλος είναι υπόλογη για την εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων. Εγώ δεν θα κρίνω, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω κατά πόσο η Ελλάδα παραβίασε οποιονδήποτε από αυτούς τους κανόνες. Θα εξετάσω πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα δημοσιεύματα που αφορούν το θέμα αυτό και γνωρίζω ότι δεν είναι μόνο ο ελληνικός λαός αλλά και ο λαός πολλών άλλων κρατών μελών έχει υποφέρει πάρα πολύ λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την ε, παραλίγο κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Ξέρω ότι ήταν ιδιαίτερο δυνηρό αυτό για πάρα πολλούς ε, πολίτες στην Ευρώπη. Ε, η διέξοδος από την κρίση είναι πολύ οδυνερή και πάνω από ε, το 50% των νέων ανθρώπων είναι ακόμα άνεργοι. Αλλά αυτό ε, δεν είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι συνέπειες, φρικτές συνέπειες μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης και θα πρέπει να αποτύσσω και φορό ε, στην Ελλάδα που κάνει τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να ξεπεράσει αυτή τη φρικτή κρίση. Αυτοί που επέκριναν τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμοστούν τα μέτρα και οι πολιτικές ε, ε, ε, παραβλέπουν το τι θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαν υπάρξει αυτές οι πολιτικές δεν είναι ότι δεν μας βολεύουν οι πολιτικές λιτότητες και αν δεν είχαμε πολιτικές λιτότητες θα είχαν συμβεί όλα και θα είχαν πάει όλα καλά και θα ήταν όλα ρόδινα. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, λάθος αναπαράσταση της πραγματικότητας και νομίζω ότι πρέπει να συγχαρώ την Ελλάδα γιατί οι προσπάθειές της έχουν αρχίσει να αποφέρουν ε, καρπούς και αυτό είναι σημαντικό ε, για το λαό της Ελλάδος. Καλύτερη νομοθεσία. Καλύτερη νομοθεσία δεν σημαίνει λιγότερη νομοθεσία. Μπορεί να σημαίνει και λιγότερη, αλλά σίγουρα σημαίνει καλύτερη, τίποτα άλλο. Βλέπουμε ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η κατάσταση με ένα κανονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντί με 28 κανονισμούς σε εθνικό επίπεδο. Καλύτερη νομοθεσία λοιπόν, better regulation, δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει λιγότερα. Υπάρχουν δυνατότητες βέβαια να κάνουμε και κάποια πράγματα λιγότερα. Κάναμε προσπάθειες μέσα σε 60 χρόνια που μας έφεραν σε μια κατάσταση που ίσως να μην χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ίσως για τον επόμενο χρόνο θα ζητήσω από τους κανονισμούς, από τους επιτρόπους να μου πούνε αν υπάρχουν κανονισμοί, αν υπάρχουν ρυθμίσεις που θα μπορούσαμε να αναιρέσουμε. Ε, για να διευκολύνουμε σαν παράδειγμα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δυσκολίες να εργαστούν με όλο αυτό το διακανονιστικό πλαίσιο. Πάντως σας λέω ξεκάθαρα το ε, ε, better regulation σημαίνει απλά καλύτερο, όχι υποχρεωτικά λιγότερο. Μπορεί να σημαίνει και μεγαλύτερο σε κάποιες περιπτώσεις. Καταλαβαίνω ότι το σύντομότερο και το μικρότερο ε, σε γραφειοκρατικό επίπεδο είναι κάτι το επιθυμητό. Αλλά όταν ολοκληρώσουμε θα σας παρουσιάσω νομίζω τα βήματα προόδου που έχουμε ε, σκοπό να σημειώσουμε στον τομέα αυτό. Για τη συνθήκη και για αλλαγές στη συνθήκη, το λέω από τώρα, έχω την αίσθηση ότι και μέσω της καλύτερης νομοθεσίας, μέσα από τη συνθήκη, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά με αυτή τη συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, να εργαστούμε πάνω σε προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το 300 δις. Ε, μπορεί να το επιτρέψει η συνθήκη. Οι Ευρωπαίοι θέλουν περισσότερη δουλειά. Οι Ευρωπαίοι θέλουν μια οικονομία η οποία να αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε τις συνθήκες για να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή βέβαια. Δεν υπάρχει η αναγκαιότητα στην παρούσα φάση. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε λίγα χρόνια. Γιατί οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις οι οποίες να απαιτούν σαν παράδειγμα αλλαγές υποχρεωτικά στη συνθήκη. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε πρώτα στον τομέα τον οικονομικό, Πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρώπη να ξαναβρει την ανάπτυξη και για να το κάνουμε αυτό δεν απαιτείται η αλλαγή της συνθήκης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν τυχόν υπάρξει και αποδειχθεί μια τέτοια αλλαγή δεν θα γίνει πραγματικότητα. Τώρα για το ποιε ενέργειες ή ποιε πράξεις ε, νομοθετικές πρέπει να αποσυρθούν. Είναι πάρα πολύ νωρί, δεν μπορώ να σα απαντήσω. Χρειάζονται χρόνο οι επίτροποι και μόνο αφού μου απαντήσουν θα σας μεταφέρω τις ε, απαντήσεις αυτές με έναν τρόπο συνεκτικό, ολοκληρωμένο, ε, κάτι το οποίο όπως είπα θα επιτρέψει στους μεμονωμένους επιτρόπους να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Εγώ είμαι υπεύθυνο, όπως ε, περιγράφει ο πρώτος αντιπρόεδρος, για τη λεγόμενη Better Regulation. Αλλά κάθε επίτροπος πρέπει να είναι υπεύθυνο για better regulation αν θέλουμε να πετύχουμε. Δεν είναι ένα θέμα ενό ανθρώπου. Ο κάθε μεμονωμένο επίτροπος και ο κάθε γενικός διευθυντή τη Επιτροπής και το εννοώ αυτό πρέπει να πιστεί ότι η καλύτερη νομοθετική ρύθμιση είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνουν οι αλλαγές εκεί όπου απαιτείται κάτι τέτοιο στο μέλλον για την κίτρινη κάρτα και για τις αντιρρήσεις των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι πολύ συγκρίσιμο με τις αντιδράσεις τις οποίες είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πρωτοβουλία των Πολιτών. Νομικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάθε δικαίωμα να αντιδρά. Πολιτικά δεν ξέρω αν ήταν πάντα σοφό το να απορρίπτει κανείς τις κίτρινες κάρτες των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπαμε και θα το επαναλάβουμε ότι αν υπάρχει ένα κοινοβούλιο κράτους μέλους που έχει προβλήματα με μια πρωτοβουλία και σηκώνει την κίτρινη κάρτα, τότε νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να πάει στο κοινοβούλιο αυτό και να εξηγήσει τις ενέργειές της και να λάβει υπόψη τις κριτικές που θα της ασκηθούν. Γιατί εάν τα κοινοβούλια αυτά μπαίνουν στον κόπο να εμπλακούν, τότε θα πρέπει να ανταποδώσει τη χάρη και το ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εξηγήσει τις θέσεις της επιτόπου και όχι να αντιδράσει απορριπτικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν υπάρχει μια κίτρινη κάρτα αυτόματα θα αποσύρεται η πρόταση της Επιτροπής. Όχι βέβαια. Η Επιτροπή θα πρέπει να εμπλακεί σε διάλογο με το συγκεκριμένο κοινοβούλιο ε, όταν και εφόσον ε, το προβλέψει η νομική διαδικασία. Συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρθηκα σε αυτό. Εξωτερική αντιπροσώπευση της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι στις ακροάσεις ε, κάναμε μία πρώτη συζήτηση γύρω από αυτό να πω ότι βασικός στόχος είναι οι χώρες οι οποίες είναι τμήμα της Ευρωζώνης και είναι και μέλη των διεθνών οικονομικών οργανισμών να έχουν στους οργανισμούς αυτούς συνεκτικές θέσεις. Αυτό θα είναι μια πρώτη σημαντική βελτίωση. Και το να έχει κανείς μία ενιαία φωνή σαν Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους οργανισμούς σημαίνει ότι θα έχει λιγότερο βάρος στο συλλεκτικό. Ε, δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο ισχύει, θα πρέπει κανείς να προσπαθήσει να διατηρήσει αυτά που έχει, αλλά για να γίνουν όλα αυτά και για να σταθμιστούν όλα αυτά πρέπει να έχουμε συμβατές μεταξύ μας και συνεκτικές θέσεις. Για την εσωτερική οργάνωση των κρατών μελών αυτό είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθούν τα κράτη-μέλη και οι πολίτες τους. Δεν είμαι κάποιος από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι έρχεται η αποκάλυψη ε, και το μέλλον δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Εγώ ζω σε αυτή τη χώρα, έχω ζήσει σε αυτή τη χώρα πάρα πολλές φορές και η χώρα αυτή έδειξε στο παρελθόν ότι είναι απολύτως ικανή χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις να αντιμετωπίζει θέματα εσωτερικής οργάνωσης και δεν επηρεάστηκε αρνητικά σε καμία περίπτωση η ευρωπαϊκή συνεργασία, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ νομίζω ότι σε καμία περίπτωση οι εσωτερικές εξελίξεις στις διάφορες χώρες δεν είναι απειλή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αντίθετα, ακριβώς γιατί τα σύνορα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν πρέπει να, να είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε σε αυτά πια. Τα κράτη-μέλη έχουν γίνει πιο χαλαρά σε σχέση με την οργάνωσή τους, και αυτή η χαλαρότητα, αυτή η πολλαπλότητα συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ τους. Φυσικά αυτό εκφράζεται και εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο στις 28 χώρες μέλη, αλλά δεν είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρέμβει γύρω από αυτό. Για τον κύριο Ντουιρό, για τη διαφάνεια και το ρόλο της διαφάνειας. Νομίζω ότι η κυρία Ντινόλφη αναφέρθηκε και αυτή. Νομίζω ότι συμφωνούμε σαν Επιτροπή και σαν Κοινοβούλιο για την διαδικασία η οποία αφορά τους μεμονωμένους επιτρόπους. Αν υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης, εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε διάλογο μαζί σας. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσω εδώ ότι η ευθύνη είναι του Προέδρου της Επιτροπής. Αυτός είναι ο Επίτροπος για τους Επιτρόπους του. Ο υπεύθυνο για τους Επιτρόπους του. Και αυτός θα κρίνει τα θέματα των προσωπικών συμφερόντων, των οικονομικών συμφερόντων, των οικογενειακών συμφερόντων. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση εδώ, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε αν θέλετε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον κάποιο πρόβλημα αλλά επειδή εγώ επιμένω στα της διαφάνειας, μια διαφάνεια η οποία θα πρέπει να μας βοηθήσει να πείσουμε τους εντολείς μας, τους εκλογής μας, ότι έχουμε ένα πρόγραμμα διαφανές και προωθούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και όχι τα προσωπικά συμφέροντα, έχουμε κάθε ε, λόγο να είμαστε διαφανείς. Τώρα για το μητρό των λόμπι, έχετε δίκιο. Εγώ δεν μπορώ να πιέσω όμως το Συμβούλιο να κάνει το ίδιο που κάνουμε εμείς η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφωνούν γύρω από αυτό και θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε την πεποίθησή μας αυτή και να προσπαθήσουμε να πείσουμε το Συμβούλιο να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα στα πλαίσια του συστήματος αυτού, καλύπτοντας τα συμφέροντα όλων αυτών που ε, έχουν σαν λόγο να νομοθετούν κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση λέγοντας ότι όσοι εμπλέκονται με ομάδες εργασίας, με ομάδες προετοιμασίας, νομοθετικών ρυθμίσεων κτλ. να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους σαν και αυτές του Μητρώου έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση. Κύριε Άνεμανς, να σας πω ότι μιλάτε πάρα πολύ καλά Ολλανδικά. Αυτό το έχουμε κοινό λοιπόν. Όλοι στο κοινοβούλιο εδώ βρίσκονται στο κοινοβούλιο γιατί υπάρχουν εκλογείς που τον ψήφισαν, ε, την ψήφισαν. Και αυτό έγινε βάσει ενός προγράμματος. Εγώ έχω άλλες ε, ιδέες λόγω του πολιτικού μου υποβάθρου και εσείς το ίδιο, αλλά δεν ε, έχουν πιο μεγάλη αξία οι δικέ μου οι ιδεολογίες από τη δική σας. Γιατί και εγώ εκλογής εκπροσωπώ και εγώ το ίδιο. Και εσείς το ίδιο. Δεν θα θεωρήσω ότι ο ένας έχει πιο πολύ βάρος από ότι ο άλλος. Ούτε πιστεύω ότι η διχοτομία που παρουσιάζετε εσείς ε, μεταξύ φεντεραλιστών και συμφερδελιστών αποτυπώνει σωστά όλες τις ιδεολογίες που εκπροσωπούνται εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλαγές και διαφορές μεταξύ κράτους μέλος, διαφορές μεταξύ, μελών, ε, διαφορές μεταξύ πολιτικού φάσματος και όλη αυτή η ποικιλομορφία νομίζω ότι φροντίζει για την πρόοδο του Κοινοβουλίου. Δεν ε, έχω όμως υποχρέωση να σκεφτώ για σας, ούτε και εσείς για μένα. Λέτε ότι είμαστε φεντεραλιστές και ότι πατάμε γκάζι σε διάφορα πράγματα. Αλλά με την απώλεια, με την ήττα στο δημοψήφισμα στη χώρα μου, αυτό που έμαθα είναι ότι όταν ε, πατάει κανείς πολύ γρήγορα γκάζι, κοιτάει πίσω του σε κάποια φάση και βλέπει ότι έχει χάσει το εκλογικό του σώμα, το λαό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει μέσα σε όλα αυτά που κάνουμε να φροντίζουμε η απόσταση μεταξύ ημών και των πολιτών μας να είναι η μικρότερη δυνατή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ρητά και ξεκάθαρα να ακούμε καλά και να εισακούμε στις επιθυμίες. Και όσοι πιστεύουν άλλα πράγματα από ότι εγώ, όπως ο κύριος Άνεμανς, όπως ε, άλλα άτομα, σε ό,τι αφορά την ε, διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις λοιπόν, αλλά ας αφήσουμε να υπάρξει αυτή η πολυμορφία για να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ μόνο και των πολιτών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, έχουμε ε, έξι λεπτά στη διάθεσή μας. τέσσερι συνάδελφοι είναι στην, στην κατάλογο των ομιλητών. Αν συμφωνήσετε να πάρετε το λόγο για ένα λεπτό, μπορείτε να πάρετε όλοι το λόγο. Ο κύριος Πλένκοβιτς είναι ο πρώτος. Μπορείτε όμως να μιλήσετε μόνο ένα λεπτό. Μην ανησυχείτε. Δεν θα μιλήσω πιο πολύ από το ένα λεπτό που μου δίνετε. Θα ήθελα να... Με ακούει και ο πρώτος αντιπρόεδρος να βάλει τα ακουστικά του. Σας συγχαίρω λοιπόν για, την, ε, το διορισμό σα. Μετά από αυτά που είπε ο κ. Σόπφλιν για τις ε, μνήμε και την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωση, Πριν από κάποιους ε, μήνε, γράψαμε στον κύριο Γιούγκερ ως μέλλον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιστολής και θα γράψουμε και προς όλους όσους τους ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα ανακοινώθηκε η εξαγωγή δημοψηφίσματο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πείτε μα ποια είναι η άποψή σα. Η άποψή σα για την ελευθερία μετακίνηση, που είναι από τα πιο ακαθόδη ζητήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, από ό,τι φαίνεται. Πιστεύετε ότι πρόκειται για ένα βήμα προ τα Εμπρό ή για ένα βήμα προ τα πίσω στην ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Σα Ευχαριστώ πολύ, Λί Πρόεδρο. Ένα λεπτό τώρα, ο κ. Πλέιρα. Com ehm, certeza. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά την συνθήκη της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα στις κρίσιμες στιγμές παρακολουθούσε στενά την κατάσταση και πάλι θα έχει καθοριστικό ρόλο λοιπόν την επόμενη, της όταν θα ψηφιστεί το σχέδιο το επενδυτικό η Επιτροπή και εσείς κυρία Αντιπρόεδρε γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων θα πρέπει να συμμετάσχει. Ελπίζω τουλάχιστον να το ξέρετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Βίβια Ρέντινγκ, ένα λεπτό. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα αυτά που είπατε για την πρωτοβουλία των πολιτών. Και σωστό είναι να γίνει μια συζήτηση Ακόμα και αν νομικός πώς έχει απορριφθεί. Αλλά μήπως θα ήταν καλύτερο να μεταρρυθμιστεί η όλη διαδικασία. Δεύτερη ερώτηση. Άκουσα τι είπατε για το κράτος δικαίου και για το σχετικό μηχανισμό στην ακρόασή σα και ότι δεν θα διστάσατε να το βάλετε σε εφαρμογή το μηχανισμό αυτό. Τι θα κάνετε όμως αν υπάρξει συστηματικό πρόβλημα στο περιθώριο του κράτους δικαίου, αν υπάρξει μια χώρα η οποία πραγματικά ζορίζει στο έπακρον τα όρια του νομικού αλλά πολιτικά μη αποδεκτού. Θα παρέμβετε και στην περίπτωση αυτή και τρίτο στοιχείο. Έχετε σκεφτεί τι θα μπορούσε να γίνει με το άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το οποίο λογικά πάντα προβάλλεται όταν τα κράτη-μέλη ξεφεύγουν από τους βασικούς ε, κανόνες ε, και τις ελευθερίες του χάρτη. Ο Ραμον Χορέγη, τελευταίος, για το τελευταίο λεπτό. Κύριε Τίμερμανς, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη βιώνει κατά πάσα πιθανότητα την πιο κρίσιμη στιγμή της ε, συναρπαστικής της ιστορίας το 74% των νέων κάτω των 24 ετών δεν ψήφισε. Να σας υπενθυμίσω μόνο αυτό το στοιχείο. Θα μπορούσαμε να σας πούμε και πολύ περισσότερα. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ σοβαρή στιγμή, κύριε Τίμερμαντς, και πραγματικά θα ήθελα να σας δώσω δύο συμβουλές. Επιτρέψτε μου το θάρρος, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν καταπηγόντως. Καταρχάς, να αναλάβει τα ενία της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης. Ούτε ο Ντράγκη, ούτε η Τρόικα, ούτε το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια οικονομική πολιτική για την Ευρώπη, ώστε ο κόσμος να δει ότι υπάρχει ε, οικονομική πολιτική και θα διαφύγουμε και τις κρίσεις. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια για το σχέδιο ολοκλήρωση τη Ένωση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν φωνέ. Ακούστηκαν και εδώ. Ορισμένε φορέ φωνάζουν και πολύ δυνατά στην Ολομέλεια κατά του ευρωπαϊκού οικοδομήματο. Αλλά υπάρχει μια πλειοψηφία. Η πλειοψηφία που υποστηρίζει αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Τίμερμαν. Υπάρχει μια πολιτική πλειοψηφία των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων που θέλουν να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν προχωρήσει, οπισθοδρομούμε. Η ε, η ευρωπαϊκή κοινωνία χρειάζεται αυτά τα δύο σημάδια ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματικά το μήνυμα ότι θα βγούμε από την κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Τίμερμανς. Ε, ε, το ερώτημα για το πιθανό δημοψήφισμα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς και αυτό επαφίεται στους Βρετανούς πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι φυλακή. Νομίζω ότι μία από τις καινοτομίες στη συνθήκη της Λισαβόνας είναι ότι ο καθής έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το επιθυμεί. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι ε, πραγματικά ε, θα με λυπήσει ιδιαίτερα εάν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θεωρώ ότι προφανώς θα είναι κακό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μπορεί να μην είναι και δική μου δουλειά να έχω άποψη από αυτού. Εάν με ρωτήσετε, θεωρώ ότι θα είναι κακό και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα το αποφασίσουν βέβαια οι Βρετανοί. Κατ' εμέ, ε, σίγουρα θα αποδυναμώσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο θα αποδυναμώσει και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσή μας με άλλες ε, παγκόσμιες δυνάμεις σε θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες και δεν είμαι βέβαιος ότι η διαπραγματευτική μας θέση θα βελτιωθεί και για το Ενωμένο Βασίλειο, εάν χρειαστεί να διαπραγματεύεται μόνο του. Ε, σας τα λέω έτσι λίγο απλά. Το θέμα της ελευθερίας ε, κυκλοφορίας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ακρογωνία λήθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς ελευθερία κυκλοφορίας πολύ δύσκολο μπορεί να έχει κάποιος ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να ε, αγνοούμε το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένες φορές έχει ε, κάποιες παράπλευρες συνέπειες για τα κράτη-μέλη, κυρίως όσον αφορά το κοινωνικό σύστημα. Έτσι είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη αν πιστεύουμε πραγματικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και τη χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, γιατί χωρίς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν θα καταφέρουμε να έχουμε την όθηση που θέλουμε για να βοηθήσουμε τους νέους Ευρωπαίους να βρουν Πρέπει να εκβιομηχανίσουμε εκ νέου την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δεξιότητες για να γίνει αυτό. Και αν ο λαός πιστεύει στα κράτη-μέλη ότι εάν υπάρχει ευρωπαϊκή κλίμακα, αν υπάρχει αυτή η αγορά, είναι τμήμα της καθημερινότητές τους, του κοινωνικού του συστήματος, ε, του, το δίκτυ ασφαλεία στι εθνικές του συνθήκε, δεν θα υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν θα υποστηρίξουν αυτό που θέλουμε εσείς και εγώ, δηλαδή ε, μια πιο ζωηρή, πιο δραστήρια Ευρώπη στο θέμα αυτό. Επομένως υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσουμε μια ψευδή διχοτόμηση μεταξύ αυτών που πιστεύουν στην ελευθερία κυκλοφορία και αυτοί που πιστεύουν ότι η ελευθερία κυκλοφορία έχει πολλές αρνητικές συνέπειες θεωρώ ότι τη χρειαζόμαστε απολύτω. Είναι ο ακρογωνιών μα λήθο. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε χωρί ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και ανοιχτοί για το γεγονό ότι πρέπει κάποιε φορέ να αντιμετωπίσουμε και τι αρνητικέ συνέπειε, ιδίω για τα κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι πρωτίστω εθνική ευθύνη, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι προετοιμασμένη να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και να μπορέσουν να επιλύσουν ε, τυχόν προβλήματα. Όσον αφορά αυτό το πακέτο των 300 ε, δισεκατομμυρίων, βεβαίως και θα συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γεννήθηκε ε, μέσω διαλόγου του Προέδρου Γιούνκερ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Ρέντινγκ μου με ρώτησε εάν πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την όλη πρωτοβουλία για τους ε, πολίτες, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ε, θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα προβλέπει η αλλαγή της συνθήκης και όπως σας είπα μόλις προηγουμένως δεν προβλέπεται αλλαγή της ε, συνθήκης. Ε, ε, υπάρχει κανονισμός για την πρωτοβουλία, αλλά δεν περιλαμβάνεται στη συνθήκη κάτι τέτοιο. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω έτσι εν θερμό. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που θέσατε και θα ήθελα να την εξετάσω. Ε, θα επανέλθω λοιπόν στο θέμα αυτό και επαναλαμβάνω ότι ακόμα και με αυτόν τον κανονισμό και πάλι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον πολιτικό διάλογο αν οι πολίτες μπουν στον κόπο να θίξουν ένα θέμα βάσει της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Το κράτος δικαίου. Άρθρο 51. παρακολούθησα τις πολύ επίκαιρε πολιτικές συζητήσεις για κάποια κρατημέλη, για όλα όσα συμβαίνουν και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά. Η θέση μου είναι η εξής. Θέλω να χρησιμοποιήσω κάθε ευκαιρία διαλόγου ως Επίτροπος με τα κράτη-μέλη εάν υπάρχουν δεδηλωμένα προβλήματα σε μια περιοχή. Και θεωρώ, κυρία Ρέντινγκ, ότι ορισμένες φορές υπάρχουν αποχρώσεις ακριβώς διότι η εκδήλωση του προβλήματος δεν παραβιάζει συγκεκριμένους κανόνες, αλλά είναι εναντίον του πνεύματος αυτού που εμείς θεωρούμε ως ευρωπαϊκά πρότυπα. Και ναι, αυτό σίγουρα θα συζητηθεί. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα διάλογο. Δεν είναι χρήσιμο να αρχίσει ο ένας να φωνάζει στον άλλον ε, το κάθε κράτος μέλος το άλλο στο δημόσιο χώρο γιατί αυτό δεν θα μας οδηγήσει σε αλλαγές. Εγώ πιστεύω σε ένα διαρθρωμένο διάλογο επί τη βάση διεξοδικής ε, ανάλυσης συγκεκριμένων ζητημάτων. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα ζητήματα, τη δυνατότητα να αντιδράσουν και ίσως να επιλύσουν τα προβλήματα. Αν όλα τα υπόλοιπα αποτύχουν, τότε ε, θα χρησιμοποιήσουμε και το άρθρο 51 και το άρθρο 37 της Ευρωπαϊκής Ένωση από εκεί πέρα, εάν χρειαστεί. Και τέλος. Ναι, υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς στις ευρωεκλογέ σε πολλά κράτη-μέλη, ελάχιστοι μπαίνουν στον κόπο να πάνε να ψηφίσουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Κοινωνία στο σύνολό τη. Δεν είναι το πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο. Και υπάρχει αυτή η ευκαιρία και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επόμενη πενταετία να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε λίγο το χάσμα, να προσεγγίσουν λίγο οι άνθρωποι αυτό που κάνουμε και θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που δουλεύουμε. Αυτό σας το λέω ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι 100% σύμφωνος με τον Ζαν κλοντ Juncker που λέει ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία για την επόμενη πενταετία. Μπορεί να μην έχουμε ούτε καν πέντε χρόνια πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που έχουν σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες βραχυπρόθεσμα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσουμε νέα κίνηση στην οικονομία, θα έχουν θέσει εργασία οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, και σίγουρα αυτό θα χρειαστεί περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε κάποιου τομεί. Αλλά θα χρειαστεί και περισσότερη ε, περισσότερο έλεγχο από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάποια περίγματα που πολύ ωραία θα ήταν να τα έχουμε, αλλά ε, δεν ε, θα ήταν ε, τόσο σημαντικά, όπω είπε και ο πρόεδρο Γιούνκερ στο Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ που ήρθατε. Χαρήκαμε που ήρθατε λοιπόν εδώ μαζί σα και θα σα καλούμε πολύ τακτικά και με χαρά μου μπορώ να σας πω ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να έρθετε να μας μιλήσετε, δεν χρειάζεται να είσαστε προσκαλεσμένος. Πολύ ορίζουμε αυτή τη στάση ανοιχτού διαλόγου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μιας και υπάρχει ακόμα η παράδοση, να σας χειροκροτήσουμε.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 Sorry, those of you who have to leave, please. Όσοι θέλετε να φύγετε, παρακαλώ, ήσυχα. Γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε την ημερήσια διάταξη και τη συνεδρίαση. Και έχω τις ανακοινώσεις που είναι σημαντικές για τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Θα πρέπει να ενημερώσω την Επιτροπή για τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση των συντονιστών, σε δύο συνεδριάσεις συντονιστών Όσοι θέλουν λοιπόν να ακούσουν τι ανακοινώσει αυτές, παρακαλώ. Στις 6 Οκτωβρίου λοιπόν ε, λάβαμε αποφάσει για τις εξή εκθεσει. Αποφασίσαμε οι συντονιστέ να υπάρχει εφαρμοστική έκθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Ελκ είναι ο για τις ε, εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας ελήφθη σε απόφαση να υπάρξει έκθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας των κτηρίων βάση της συνθήκης της Λισαβόνας βάση της εφιστάμενης συνθήκης Έλμας Μπρόκ ε, από τους σοσιαλιστές έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, για την ε, σύσταση και την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Άλντε Γκίβερ Χόφστα, το εισηγητής. Απόφαση για την νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση των συνθήκων για την ενιαία έδρα, τη μία και μοναδική έδρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση αυτή πάει στο ECR. Έκθεση ίδια πρωτοβουλία για τις θεσμικέ επιπτώσει του νέου μηχανισμού οικονομικής διακυβέρνησης. Πώ θα βελτιωθεί η δημοκρατική Λογοδοσία. Έκθεση που προτάθηκε από την ΚΟΗ. Ο κύριος Κατρούγκαλος θα είναι εισηγητής. Συμφωνήσαμε ο Γραμμόν Κουρανέγκη να διοριστεί από τους σοσιαλιστές ως ο νέος εισηγητής που θα αντικαταστήσει τον Ντέιβιντ Μάρτιν για την έκθεση για, την, για τα δικαιώματα υποβολής ερωτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένουμε θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου επίσης συμφωνήσαμε για την έκθεση για την αναθεώρηση του εκλογικού δικαίου νομοθετικής ε, φύσης έκθεσης δύο εισηγητές από το ΕΛΚ και από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Αποφασίσαμε επίσης στις 6 Οκτωβρίου για τις ακροάσεις και τις επιτροπές. Σε ό,τι αφορά τις ακροάσεις ε, θα γίνουν ακροάσεις για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αρχές ε, του επόμενου έτους ακρόαση για τις θεσμικές επιπτώσεις του νέου μηχανισμού οικονομικής διακυβέρνησης και το ρόλο του Eurogroup για το πώς θα βελτιωθεί η δημοκρατική λογοθεσία σε συνεργασία με την Επιτροπή ΕΚΟΝ και αυτό επίσης θα είναι την άνοιξη του 2015, Μάρτιο ή Απρίλιο. Επίσης, ακροάσεις για το θεσμικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του πλαισίου του, των συνθήκων και πέρα από τις εφιστάμενες συνθήκες θα, λάβει χώρα, λάβουν χώρα Απρίλιο ή Μάιο, θα αποτελέσουν και συνέχεια του εργαστηρίου που είχαμε σήμερα. Επίσης, συμφωνήσαμε για τις μήνυα σε ε, λίγο πιο μικρές ε, σε έκταση σε ό,τι αφορά την προσχώρηση στον Ευρωπαϊκό, στο ECHR και σε ό,τι αφορά την ε, προσχώρηση στον Ευρωπαϊκό χάρτη σε ό,τι αφορά τις αποστολές εκτός των τριών ε, εδρών εργασίας. Θα ζητήσουμε από τη διάσκεψη των Προέδρων να υπάρξει αποστολή στη Ρήγα το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο σε ό,τι αφορά την ε, πρωτοβουλία της χώρας και στο Βερολίνο τον Ιούνιο του 2015. Στο δεύτερο ήμιση θα έχουμε επίσκεψη στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον. Σήμερα στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών συμφωνήσαμε να δώσουμε την γνωμοδότηση για τον κανονισμό για τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα, όπου και συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων με καθήλυνη αρμόδια την ΛΥΜΠΕ. Ο κ. Σόλτς θα είναι ο εισήγητης εξ όσων κατάλαβα. Συμφωνήσαμε επίσης για την έκθεση που προτείνουν οι πράσινοι. Δεν έχω τον τίτλο «Διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατία». Συμφωνήσαμε για την έκθεση, αλλά η τελική απόφαση αναβλήθηκε μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών, στο ιστορικό των πολιτικών εβδομάδων. Σχέδιο ψηφίσματος της κυρίας Μπιτσότο για την ε, μία και μόνη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα αυτού θα εξεταστεί στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης. Δεν σημαίνει αυτό το δικό μας ψήφισμα θα, θα συνδυαστεί με την έκθεση νομοθετικού περιεχομένου. Επίσης, συμφωνήσαμε για τη σύνθεση της ομάδας εργασίας για τον κανονισμό. Δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα εργασίας στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου και σήμερα συμφωνήσαμε ότι θα καλέσουμε και ένα μη εγγυγραμμένο να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις ως παρατηρητής. Αυτά συμφώνησαν λοιπόν οι συντονιστές σήμερα και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα εγκριθούν οι αποφάσεις αυτές. Δεν βλέπω να υπάρχουν ενστάσεις και άρα περνάω στο 4 το οποίο είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης το οποίο το κάναμε το πρωί Ιουλίου και Σεπτεμβρίου τα έχετε στη διάθεσή σας και ως ήθισε θεωρούνται εγκεκριμένα αν δεν έχει εκφραστεί ένσταση μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης. Αυτά σε ό,τι αφορά τα της Επιτροπής μας. Και τώρα να περάσω και πάλι στο μεγάλο θέμα, το σημερινό το εργαστήρι μας και συζητήσεις μας για τις ε, προκλήσεις στον τομέα των σταγματικών υποθέσεων στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Και τώρα περνάμε πλέον στη συνεδρίαση που έχει αφιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Τρίτο πάνελ σήμερα και να ξεκινήσουμε με το Πανεπιστήμιο της Πίζα και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα της Φλωρεντίας. Ο προσκεκλημένος μας ε, θα είναι ο πρώτος ομιλητής, ομιλητής για την δομή του συστήματος της Ευρώπης μετά τις εκλογές του 2014. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μία παρουσίαση PowerPoint. Okay. All right. Thanks. Um, actually, uh, this presentation is the, on the evolution of the Euro Party system αφορά τις εξελίξεις των ελεγωμένων ευρωπαϊκών κομμάτων. Γιατί δεν χρειάζεται να δώσω πολλές εξηγήσεις σε αυτό. Νομίζω ότι όλοι εδώ είμαι πεπισμένος ότι γνωρίζουν ότι το δημοκρατικό έλλειμμα και το πρόβλημα του δημοκρατικού έλλειμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σοβαρό. όπως ακούσαμε και από τους προηγούμενους ομιλητές, πόσο μάλλον που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τώρα πλέον περισσότερες αρμοδιότητες. Εγώ συγκεντρώνω την προσοχή μου στις ευρωπαϊκές εκλογές γιατί πιστεύετε τότε, όταν άρχισαν να διεξάγονται, ότι θα γινόταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο ισχυρό θα ήταν σε θέση να επιλέξει ανάμεσα σε εναλλακτικές πολιτικές λύσεις και θα γινόταν γενικά πιο πολιτικοποιημένο. Αυτό δεν έγινε ακόμα, έτσι νομίζω εγώ. Αυτό που ονομάζουμε κανονικές δημοκρατίες εισαγωγικά. Τι σημαίνει αυτό. Τα κόμματα παίζουν αυτό το ρόλο με ένα κεντρικό σύστημα, ένα κοινό κομματικό σύστημα. Εμείς πιστεύουμε ότι όσο ε, πιο θεσμικά και διαρθρωμένα είναι τα κομματικά συστήματα τόσο το καλύτερο. Συνίσταται από δύο βασικά συστατικά, τις ενότητες και τη δομή. Οι ενότητες είναι τα κόμματα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια ιδέα του πώς είναι ακριβώς ε, οι ενότητες, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε το σύστημα στο σύνολό του και στη δομή του. Η ύπαρξη του κομματικού συστήματος μπορεί να θεωρηθεί σαν προϋπόθεση για τη δημοκρατία. Λόγοι είναι οι εξής. επηρεάζει το κομματικό σύστημα την έννοια της αντιπροσωπευτικότητας, τη σταθερότητα της κυβέρνησης, της επιδόσεις της κυβέρνησης και την νομιμοποίηση των κυβερνητικών εισφορών. Έτσι εμφανίζεται το σύστημα στα διάφορα κράτη-μέλη και έτσι θα έπρεπε να εμφανίζεται για πολλούς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ερχόμαστε τώρα στις εκλογές του 2014. Στόχος αυτής της παρουσίασης, κεντρικός στόχος, είναι να ελέγξει τις επιπτώσεις των εκλογών αυτών που είχαν κάποια διάσταση επαναστατική, θα έλεγε κανείς, στο ευρωπαϊκό κομματικό σύστημα και στον ρόλο προώθησης της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. θα δούμε με γενικό τρόπο τις ενότητες, τα κόμματα δηλαδή, και με πιο ειδικό τρόπο την δομή τους, την οργάνωσή τους. Εμείς θα εξετάσουμε λίγο και την συμπεριληπτικότητα των κομμάτων. Όσο πιο υψηλή είναι, τόσο το καλύτερο τα κόμματα με υψηλό τέτοιο επίπεδο είναι πιο ε, διεθνικά θα έλεγα. Για να μπορεί ένα κόμμα να εργάζεται σωστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι ένα πραγματικά ευρωπαϊκό κόμμα στο εσωτερικό της δομής του. Το άλλο πράγμα που καλούμεθα να εξετάσουμε είναι η εξάρτηση των κομμάτων αυτών από τις μεγάλες τους εθνικές αντιπροσωπίες. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε το αντίθετο, ότι όσο πιο χαμηλή είναι η εξάρτηση αυτή, τόσο το καλύτερο. Γιατί, Γιατί απλά πιστεύουμε ότι μια μεγάλη εθνική αντιπροσωπεία θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην διεθνοποίηση. Και γι' αυτό ακριβώς η κυρίαρχη πανεπιστημιακή αντίληψη είναι ότι αν υπάρχουν ε, μεγάλες ε, εθνικές αντιπροσωπείες, τότε οι αντιστάσεις θα είναι υψηλές. Εδώ θα σας δώσω κάποια επιπλέον στοιχεία. Είναι τα δεδομένα τα οποία συλλέξαμε σχετικά με την δυνατότητα συμπερίληψης που έχουν οι πολιτικές ομάδες των κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η εξάρτησή τους από τις μεγάλες εθνικές αντιπροσωπείες. Στις πρόσθετες έξι στήλες σας δίνουν στοιχεία συμπεριληπτικότητας όπως είπαμε και ταυτόχρονα έχουμε τα στοιχεία του 2009 και του 2014 τα οποία καλύπτουν τα ποσοστά των μεγαλύτερων συνιστοσών εθνικών μέσα στο κόμμα. Μέσα στην ομάδα καλύτερα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές και οι Φιλελεύθεροι ιστορικά ήταν πάρα πολύ πάντα συμπεριληπτική, κάλυπταν δηλαδή ε, σε υψηλό επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο και αναφέρομαι σε απόψεις πανεπιστημιακού τύπου, δεν κάνω πολιτική παρουσία, σε θεωρείται ο πυρήνα στα τρία αυτά κόμματα της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα επόμενα κόμματα η ΚΟΕ, η πράσινη και τώρα πλέον και η συντηρητική είναι σε μια ενδιάμεση κατηγορία. Δεν είναι διεθνικά, αλλά είναι πολυεθνικά και αυτά. Έχουν εκπροσώπους από αρκετές χώρες, όχι όλες από αρκετές χώρες όμως. Αυτό θεωρείται ένα υψηλό επίτευγμα γιατί σε πάρα πολλές χώρες το να φτάσει κανείς και να αποκτήσει μία έδρα είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν αποστέλουν πάνω από έξι ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά. Και τέλος, στην τελευταία κατηγορία, έχουμε το EFD και τα λοιπά, με 7 στους 28. 7 δηλαδή εθνικές αντιπροσωπείες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο για την ίδια την πολιτική ομάδα και την επιβίωση αυτής της ομάδας. Είδαμε ότι τον προηγούμενο μήνα υπήρξαν προβλήματα, αλλά για μια ακόμη φορά, και εδώ κάνω μια ακαδημαϊκού τύπου ανάλυση, δεν θέλω να θίξω κανένα, είναι ένα δυνητικό πρόβλημα και για το σύστημα το πολιτικό στο σύνολό του. Είναι μια πιθανή πηγή αστάθειας το να έχει μια πολιτική ομάδα η οποία εκπροσωπεί κόμματα εθνικά και η οποία να είναι πάντα έτοιμη προς κατάρρευση. Ας δούμε τώρα τις μεγάλες συνιστώσεις. Βλέπετε ότι οι τρεις πρώτες μεγάλες πολιτικές ομάδες δεν εξαρτώνται πραγματικά από μια μεμονωμένη εθνική αντιπροσωπεία. 15%, 11%, 16%, 14%. Αυτά είναι χαμηλά ποσοστά. Μετά έχουμε στις επόμενες ομάδες μια ενδιάμεση κατάσταση και το καλοδεχούμενο μετά τις εκλογές του 2014, στα αποτελέσματα δηλαδή, είναι ότι οι συντηρητικοί τώρα έχουν την μεγαλύτερη εθνική αντιπροσωπεία 26%, 28,6%. Όταν το πω αυτό μπορεί κάποιοι να μην τους αρέσει από το ECR, αλλά δυνητικά και αυτοί προχωρούν στη λεγόμενη διεθνοποίηση. Η FD είναι, θα έλεγα, αυτό που ονομάζουμε μονοκομματική ομάδα. Δεν υπάρχουν βέβαια ακόμα μονοκομματικές ομάδες, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν. Αλλά όταν μια αντιπροσωπεία έχει το 50% των μελών μιας πολιτικής ομάδας, τότε μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η εθνική αυτή αντιπροσωπεία θα λειτουργεί με αυτόνομο τρόπο. Οπότε όσο μεγαλύτερη είναι ποσοστιαία η συμμετοχή ενός κόμματος, τόσο περισσότερο θα συμπεριφέρεται σαν ενίο κόμμα. Δεν αναφέρομαι τώρα στην πρακτική τελευταία, αλλά στο παρελθόν αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ο επόμενος πίνακας εξετάζει τη δομή των ευρωπαϊκών κομμάτων, αυτών καθεαυτών. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ είναι να δώσουμε κάποια μετρήσιμα μεγέθη. Απλά. Σαν παράδειγμα, ο αριθμός των ομάδων κομμάτων. Όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο. Γιατί υπάρχει μικρή διασπορά και λιγότερη αστάθεια. Οι τα επόμενα μεγέθη ε, θέλουν κάποιες εξηγήσεις. Ο αριθμός των πραγματικών κομμάτων. Αυτός είναι ένας κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ομάδων κομμάτων αλλά και, το σχετικό μέγεθος των μεγάλων. Οι πανεπιστημιακοί πιστεύουν πάντα ότι και εδώ ο χαμηλότερος είναι ο αριθμός, πως τόσο χαμηλότερος τόσο το καλύτερο. Τώρα το ποσοστό των μη εγγεγραμμένων ευρωβουλευτών είναι ένα ποσοστό το οποίο θα θέλαμε εμείς να μειούται. Αναφέρεται την αντίσταση που υπάρχει στην, ε, ε, στην απόκτηση ευρωπαϊκού χαρακτήρα των μελών ενός κόμματος. Αντίθετα, το ποσοστό των ευρωβουλευτών της λεγόμενες ε, ομάδες, τις κεντρικές, τις σημαντικές, όσο υψηλότερο είναι τόσο το καλύτερο. Εδώ βλέπετε τον πίνακα. Φαίνονται οι αριθμοί, μπορούν να διαβαστούν, δεν είναι πάρα πολύ μικροί. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι τον αριθμό των κομμάτων, των ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θεωρούμε τους μία γεγραμμένους μία ομάδα, κατ' οικονομίαν, γιατί μας διευκολύνει στην καταμέτρηση των υπολείπων δικτών. Πρόκειται για μια αυθαίρετη επιλογή. Αλλά μιας και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τάσεις, δεν αλλοιώνεται η ανάλυση. Αν δεν σας αρέσει αυτή η επιλογή, είναι θα πρέπει να μικρύνεται κάπως ε, το δείγμα. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι μια τάση και η τάση δείχνει ότι δεν έχουν υπάρξει αλλαγές από το 1979 μέχρι το 2014. Υπάρχουν κάποιες απομονωμένες ε, λεπτομέρειες αντίθετες, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο για να σταθώ σε αυτά. Όλοι οι άλλοι δείκτες όμως δείχνουν ότι στις εκλογές του 2014 ότι ήταν αυτές οι οποίες επηρέασαν περισσότερο από ποτέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν ίσως αναμενόμενο σε πολιτικό επίπεδο αλλά δεν ήταν κάτι το δεδομένο πριν από τις εκλογές. Όταν δει κανείς αυτούς τους αριθμούς, βλέπουμε ότι οδηγούν τις δομές αυτές στα επίπεδα ε, τα οποία, στα οποία είχε φτάσει το 1979 όταν εξελέγει το πρώτο κοινοβούλιο. οι δομές των κομματικών θα έλεγα εκπροσωπήσεων ήταν οι ίδιες, εκτός από τους μη εγγεγραμμένους βέβαια. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι είναι και τότε μία μεμονωμένη πολιτική ομάδα, ήταν απλά μέλη σε μία ομάδα και όχι ε, μέλη κομμάτων που ανήκαν σε μία ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, η ανάπτυξη σε επίπεδο διαφθρωτικών χαρακτηριστικών του Κοινοβουλίου έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο το 2014 και είχαμε κάποια δείγματα από το 2009 για το τι θα συνέβαινε το 2014. Δεν έχω περισσότερες διαφάνειες. Τα συμπεράσματα θα τα πω κάπως προσωπικά. Το τι θα πρέπει να περιμένει κανείς και το τι συνέβη. Τι μάλλον αναμενόταν να συμβεί και το τι συνέβη. Ένα σωστά διαφραμμένο κομματικό σύστημα είναι σημαντικό για να είναι ισχυρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτό υπάρχει μια σύγκληση απόψεων. Αλλά για το κομματικό σύστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά στα πλαίσια της ενίσχυσης της δημοκρατίας χρειάζεται να είναι ανταγωνιστικό και πολιτικοποιημένο. Αυτό το οποίο έχουμε λοιπόν εδώ είναι δύο πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν. Από τη μία θέλει κανείς να έχει τις μεγάλες πολιτικές ομάδες με πολλούς φιλελευθέρους, πολλούς ε, χριστιανοδημοκράτες και πολλούς σοσιαλιστές. Από την άλλη, εάν πράγματι θέλει κανείς να έχει ένα πραγματικά ανταγωνιστικό κόμμα, πρέπει να έχει και μια ισχυρή αντιπολίτευση, ένα καλό κομματικό σύστημα ενώ και γι' αυτό στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο είτε θα διαρθρωθεί περισσότερο, στενότερα, είτε θα είναι πιο πολιτικοποιημένο. Αυτό δεν θα το πω εγώ. Εξαρτάται κανείς από τις απόψεις τις οποίες έχει πολιτικά. Η άποψή μου λοιπόν, δευτερευόντως, και επί τη βάση της εμπειρίας που έχω, ήμουν υπεύθυνο και στην πρώτη, στον πρώτη έρευνα για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 1983. Τότε ήταν σημαντικό να στοχεύει κανείς την ισχυροποίηση των πολιτικών κομματικών ομάδων. Το Κοινοβούλιο τώρα μπορεί να είναι ίσως ε, και λιγότερο διαρθρωμένο θεσμικά, αλλά περισσότερο σίγουρα πολιτικοποιημένο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάρτη. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον ε, κύριο Μπαλόρτη για να συνεχίσει. να δω τι θα πείτε, κύριε Καρλαουζή, μεταξύ συνεργασίας και ανταγωνισμού, λέτε. Να δούμε σε τι συμπέρασμα θα καταλήξετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Το θέμα της παρουσίασής μου είναι οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών του ομάδων και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Να σας πω λίγο το διάγραμμα της παρουσίασής μου. Καταρχάς θα σας κάνω μια εισαγωγή για τις διάφορες έννοιες, μετά θα μιλήσουμε για τη σημασία της ιστορίας ε, και την ανάπτυξη αυτών των ε, ε, ευρωπαϊκών δομών. Το τρίτο τμήμα είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο, το τέταρτο φορά τη συνεργασία και στο τέλος φυσικά θα σας παρουσιάσω κάποια συμπεράσματα. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Το 1993 δύο εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί ε, πολιτικών επιστημών είπαν ότι μπορούμε να αναλύσουμε τις δομές των εθνικών πολιτικών κομμάτων ε, χωρίζοντάς τα σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Ο παρακαθήμενός μου, ο κύριος Μπάρτι, το 2006 ε, είπε ότι μπορούμε να αναλύσουμε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα χρησιμοποιώντας το ίδιο διάγραμμα. Έχουμε μία φάση που λέγεται ε, κόμμα σε δημόσια αξιώματα που είναι τα, οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε και τα πολιτικά κόμματα σε κεντρικές θέσεις που είναι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή και έχουμε και ένα τρίτο στάδιο τα κόμματα επιτόπου που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν εκπροσωπούνται από μεμονωμένα μέλη γιατί ελάχιστα πολιτικά κόμματα επιτρέπουν να είναι κάποιο ε, μέλος ε, και εκπροσωπούνται από τα διάφορα πολιτικά κόμματα σε εθνικό επίπεδο. Επομένως έχουμε τα εθνικά κόμματα. Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των τριών φάσεων μπορούν να αποκληθούν ε, ευρωπαϊκό κόμμα. Θα δούμε τι γίνεται όταν είναι ισχυρές οι σχέσεις και υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών φάσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν λειτουργεί βέβαια το διάγραμμα αυτό και εδώ ε, θα σας δείξω ένα άλλο διάγραμμα που θα μπορούμε, ε, μπορούσαμε ίσως να το αποκαλούμε το ευρωπαϊκό επίπεδο, το τέταρτο στάδιο των εθνικών κομμάτων, διότι πλέον δεν έχουμε μόνο τρεις διαφορετικές φάσεις, αλλά έχουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο ως μια φάση εξάρτησης των εθνικών κομμάτων. Είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ευρωπαϊκά κόμματα βάσει αυτού του διαγράμματος. Να πούμε δύο λόγια για την ιστορία. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επομένω φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πολύ καλά την ιστορία των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Α δούμε λίγο την ιστορία των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μια μπλε γραμμή εδώ που βλέπετε και αυτή η γραμμή είναι ο κανονισμός 2014 του 2013. Και αυτός ο κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά το 2004 και η βασική συνέπεια είναι η χρηματοδότηση. Το γεγονός ότι τα κονδύλια προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ευρωπαϊκά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέντε πολιτικές οικογένειες έχουν ήδη συστήσει πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσαμε να τα αποκαλούμε ε, διεθνικές ομοσπονδίες κομμάτων, πριν από την εισαγωγή της χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά το 2004 βέβαια συστήθηκαν πολλά άλλα πολιτικά κόμματα. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ε, ε, δύο διαφορετικών ομάδων και τα πέντε πολιτικά κόμματα τα οποία είχαν ιδρυθεί πριν από το 2004 είναι ε, ε, κόμματα τα οποία είναι υπέρ της Ευρώπης. Ενώ μετά το 2004 τα, πολλά από τα κόμματα που ιδρύθηκαν ε, μετά από αυτή την ημερομηνία έχουν ε, διαφορετικές απόψεις για τα διάφορα στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ας δούμε λίγο τι γίνεται μεταξύ του ανταγωνισμού με το, μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Έχω τρεις ε, ε, παράγοντες εδώ, τη χρηματοδότηση, ε, το προσωπικό και την πράσπιση των συνόρων. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η πράσινη γραμμή είναι τα κονδύλια τα οποία λαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ υψηλότερη από τις άλλες δύο γραμμές που είναι τα κονδύλια τα οποία λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα. Αν το δούμε και σε διάγραμμα ε, πίτας, ε, βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση μεν στο μερίδιο, αλλά η μεγαλύτερη χρηματοδότηση είναι για τις πολιτικές ομάδες. Παρά το γεγονός ότι το μερίδιο το οποίο ε, καταλαμβάνουν οι πολιτικές ομάδες στη χρηματοδότηση θα μειωθεί. Ε, οι πολιτικές ομάδες λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ισχυρότερες αλλά θα μειωθεί αυτή ο συσχετισμός δυνάμεων. Τώρα, προσωπικό. Εδώ, στην ίδια ευθεία, έχουμε πολιτικές ομάδες και πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο, το PPL e είναι αυτό, το οποίο ανήκει στην ίδια πολιτική ομάδα. Απομένως έχουμε το ΕΛΚΟΣ πολιτική ομάδα και εδώ έχουμε το προσωπικό που αριθμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ έχουμε και το ΕΛΚ ως πολιτικό κόμμα και εδώ έχουμε και το προσωπικό τους. Και εδώ έχουμε και την αναλογία μεταξύ των δύο αυτών τιμών και βλέπουμε ότι η πολιτική ομάδα είναι 4,61 φορές ισχυρότερη από το ΕΛΚ ως πολιτικό κόμμα. Και το αυτό ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, διότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ υψηλότερα από το 0. EP groups are stronger than the uh, political parties at the European level. Let's talk about the criteria. Τώρα, τα κριτήρια ίδρυσης. Έχουμε δύο είδη κριτηρίων. Ποιοτικά κριτήρια και για τις πολιτικές ομάδες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα πολιτικά κόμματα, αλλά ο έλεγχος αυτός των ποιοτικών ε, κριτηρίων δεν είναι ε, τόσο αποτελεσματική γιατί είναι όσο επιτοπλίσαν εκ των υστέρων. Δεν είναι αποτελεσματικά για να δούμε κατά πόσον συμφέρει να υπάρχει ή να ιδρύεται ένα νέο πολιτικό κόμμα ή μια πολιτική ομάδα. Ποσοτικά κριτήρια. Αυτή είναι εκ των ε, προτέρων έλεγχη και είναι πολύ πιο αποτελεσματική τα ελάχιστα κριτήρια προκειμένου να ιδρυθεί μια ομάδα. Πρέπει να έχουμε 25 ευρωβουλευτές από 7 διαφορετικές χώρες και ας δούμε τώρα και τα κριτήρια για τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κριτήρια εδώ είναι πολύ πιο χαμηλά. Χρειάζονται 7 βουλευτές, ευρωβουλευτές, εθνικοί βουλευτές, ε, ή και 7 που μπορεί να προέρχονται από περιφερειακά κοινοβούλια, από 7 διαφορετικές χώρες, μπορούν να δημιουργήσουν ένα κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, οι ομάδες είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπερασπιστούν ε, το, ε, την παρουσία τους. Μπορούν να αποφύγουν ουσιαστικά την παρουσία άλλων πολιτικών ομάδων που σημαίνει ότι θα υπάρξουν περισσότερα χρήματα για αυτούς γιατί αν υπάρξουν και νέες πολιτικές ομάδες τότε θα λάβουν και αυτή η χρηματοδότηση από τον ίδιο Κορβανά. Επομένως βλέπουμε ότι οι πολιτικές ομάδες είναι ισχυρότερες από τα πολιτικά κόμματα. Ας πάμε τώρα στην ε, συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο δομών. Εδώ έχουμε την ε, συμμετοχή την, ε, σε ένα πολιτικό κόμμα, την παρουσία των ευρωβουλευτών στις πολιτικές ομάδες και τη σχέση μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των πολιτικών κομμάτων. Τι είναι ε, ε η συμμετοχή σε ένα πολιτικό κόμμα, σε μια πολιτική ομάδα. Αυτά είναι στοιχεία από την προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από το ΕΛΚ το 2014 έχουμε ε, μέχρι το 2014 είχαμε 265 βουλευτές. Από αυτούς οι 263 ήταν μέλη εθνικών κομμάτων που συμμετείχαν στο ΕΛΚ ως κόμμα. Είναι λίγο περίπλοκο αυτό, αλλά βλέπετε εδώ ότι το ποσοστό των ευρωβουλευτών που ανήκαν στην, και στην ομάδα και στο πολιτικό κόμμα ανερχόταν στο 99,2%. Ε, τα πράγματα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ήταν λίγο διαφορετικά, γιατί από τους 184 οι 161 ήταν ε, μέλη εθνικών κομμάτων που συμμετέχουν στο κόμμα των ε, Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Επομένως το ποσοστό ήταν 88%. Και αυτό κυρίως διότι το Ιταλικό Δημοκρατικό Κόμμα τότε ήταν μέλος της ομάδος ΜΕΝ αλλά δεν συμμετείχε στο κόμμα ΔΕ. Και βλέπετε εδώ τι σημαίνει ότι να ανήκει και στο κόμμα η ομάδα. Το σκεπτικό είναι ότι όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό, τόσο ισχυρότερη είναι η σχέση. Όσον αφορά τώρα την παρουσία ε, των Ευρωβουλευτών στα όργανα του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Έχω ε, λάβει κάποια στοιχεία μόνο για τα ε, κογκρέσα και τα, ή τα συμβούλια, μπορεί να είναι ένα συμβούλιο, μια διεύθυνση ή οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά όλοι οι ευρωβουλευτές μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ή σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου στα ε, όργανα των πολιτικών ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό διαφέρει. Κάποια πολιτικά κόμματα από τα συμβούλια, σε κάποια πολιτικά κόμματα επιτρέπεται να συμμετέχει κάποιος ε, αν είναι ευρωβουλευτές ε, στο Συμβούλιο, ενώ κάποιοι άλλοι δεν επιτρέπουν στους ευρωβουλευτές να συμμετέχουν στο Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο διαφορετικών δομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι τόσο ισχυρές σε αυτή την περίπτωση. Και εδώ βλέπετε ένα τελευταίο δείχτη που μας δείχνει τις επίσημες σχέσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδα λίγο τα καταστατικά των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν δείτε το καταστατικό του ΕΛΚ, εκεί λέγεται ότι υπάρχει επίσημη συνεργασία με την πολιτική ομάδα. Το αυτό ισχύει και για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Είναι επίσημη η σχέση μεταξύ της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών όπως επίσης και για τους φιλελευθέρους και για τους πρασίνους και το καθεξής. Τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, τα τρία τελευταία, δεν έχουν επίσημες σχέσεις. Το ECPM, το EAF και το MELT δεν έχουν κάποια επίσημη σχέση με τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Conclusions. Uh, e Τελευταίες παρατηρήσεις. Οι πολιτικές ομάδες είναι ισχυρότερες από τα ευρωπαϊκά κόμματα παρά το γεγονό ότι μειώνεται αυτή η ισχύ. Σε γενικές γραμμές οι ισχυρότερε σχέσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών κομμάτων υπάρχουν για τα κράτη τα οποία ιδρύθη, για τα κόμματα συγγνώμη, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από το 2004, δηλαδή τα λεγόμενα κόμματα που είναι υπέρ τη Ευρώπη. Και τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα ε, που δημιουργήθηκαν μετά το 2004 δεν έχουν ε, τέτοιες ε, σχέσεις. Από τα τρία αυτά μοντέλα θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να αναλύσουμε τις δομές οι οποίες ιδρύθηκαν πριν από το 2004, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, αυτή την τέταρτη φάση, είναι χρήσιμο να αναλύσουμε δομές οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά το 2004. Τώρα και μια σύσταση για τους ακαδημαϊκούς. Μην θεωρείτε ε, πλέον ότι τα κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν πριν από το 2004 αποτελούν πρότυπο για τα άλλα κόμματα, διότι πολλά από αυτά τα νέα κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν μετά το 2004 δεν θέλουν να μετατρέψουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία σε μια συνηθισμένη, σε μια ομαλή δημοκρατία, όπως είναι η δημοκρατία μιας ε, χώρας. Και για τους υπολείπους. Εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα. Το άρθρο 491 της συνθήκης του Μάστρικ εισήγαγε το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντικά για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί συνεισφέρουν στην εξοικείωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δεύτερο είναι ότι εκφράζουν την πολιτική βούληση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται όμως όταν η πολιτική βούληση των πολιτών της Ένωσης είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι για πάρα πολλά χρόνια το μόνο που φροντίζαμε εμείς ως ε, ακαδημαϊκοί και πρακτικοί ήταν ε, το πρώτο τμήμα του άρθρου, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο τμήμα. Εγώ λοιπόν θεωρώ να μην, ότι ε, δεν θα πρέπει να θεωρούμε τα κόμματα τα οποία είναι αντιευρωπαϊστές ε, ο, ότι δεν είναι ευρωπαϊκά, γιατί και αυτοί ε, νομιμοποιούνται ε, για το θέμα της ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και τώρα θα περάσουμε στην κυρία Μάρτα Μπαλιστέρος για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών και είσαστε εμπειρογνώμονας και εργάζεστε επί της πρακτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας αυτής. Πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό, γιατί όπως ξέρετε προσεγγίζει και η φάση της αναθεώρησης ε, της πρωτοβουλίας. Thank you very much for giving... Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ την ευκαιρία για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της ε, μελέτης. Είμαι Ισπανίδα δικηγόρος και εργάστηκα επί 22 χρόνια στις Βρυξέλλες για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που άπτονται κυρίως ε, του περιβαλλοντικού δικαίου. Εργάζομαι στην εταιρεία Milieu που είναι συμβουλευτική εταιρεία και παρέχει συμβουλές ε, σε δημόσια όργανα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ήμασταν υπεύθυνοι για την ανάπτυξη μιας μελέτης για να συζητήσουμε και να αναλύσουμε αυτά που έγιναν για να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την πρώτη περίοδο. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε μάλλον η πρωτοβουλία των πολιτών από τη συνθήκη της Λισαβόνας προκειμένου να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψη αποφάσεων της ευρωπαϊκή Ένωσης. Το Κοινοβούλιο ήθελε να κατανοήσει κατά πόσον τα διάφορα κριτήρια τα οποία οι διάφορε απαιτήσει οι οποίοι τέθηκαν στο άρθρο 11 ένα εκατομμύριο δηλαδή πολίτες από 7 κράτη-μέλη ή το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών περιορίζεται στο να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πράξη, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο αυτό το πράξει ή όχι. Ή οποιαδήποτε άλλη, οποιοδήποτε άλλος όρος ο οποίος στήφεται από το άρθρο 211 του 2011 ότι είναι υπερβολικά αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει πραγματικά να ζητηθεί η πρωτοβουλία των πολιτών. Ο λόγος λοιπόν για τη διεξαγωγή της μελέτης ήταν για να δούμε κατά πόσο πρόκειτο για ένα αποτελεσματικό μέσο για την πρόθεση της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ήταν αρκετά δημοκρατικό ως μέσο. Είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον θα προβεί σε νομοθετική πράξη. Αξίζει ο κόπος να συλλεχθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές. Είναι πάρα πολλές. Είναι πολύ περιοριστικό το γεγονός ότι προβλέπεται ένα έτος. Όλα αυτά λοιπόν μας ζητήθηκε να τα ερευνήσουμε. Ο λόγος για τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία ήταν ο εξής. Όταν έγινε η μελέτη από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάιο του 14. έγιναν 46 πρωτοβουλίες. Μόνο 28 εξ αυτών καταγράφηκαν και εξ αυτών δύο μόνο ήταν επιτυχείς ως πρωτοβουλίες, δηλαδή έφτασαν το φράγμα του ενός εκατομμυρίου. Ξέρω ότι υπάρχει κι άλλη μία τώρα και υπήρξαν δύο απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν έγινε πρόταση νομοθετικής πράξης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγιναν λοιπόν εξηγήσει, δόθηκαν εξηγήσει για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν υπήρξε τελικά πρόταση νομοθετική πράξη. Αυτό περιμέναμε από την πρωτοβουλία. Αυτό ήταν το αντικείμενο της ανάλυσης της έρευνάς μας. Μας ζήτησαν να βρούμε τα εμπόδια για τους διοργανωτές. Ενδεχόμενες λύσεις, είτε από τη βιβλιογραφία είτε από τις συζητήσεις μαζί με τους διοργανωτές. Η μεθοδολογία μας λοιπόν ήταν η εξή. Συζητήσαμε με τους διοργανωτές, με τις εθνικές αρχές που εμπλέκονται κάποιους εκπροσώπους, εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων ε, βουλευτών από τρει, τρεις ομάδες, το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεων. Κάναμε και σχετική έρευνα χρησιμοποίησαμε ένα πάνελ από εμπειρογνώμονες για να επαληθεύσουμε τη μεθοδολογία μας. Νομίζω ότι πιο πολλοί ε, από εσάς γνωρίζετε ποια είναι η διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Δεν πρόκειται να την αναλύσω. Ένα σημείο θέλω να τονίσω. Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών να καταγραφεί, γίνεται ένας πρώτος έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και ελέγχει κατά πόσον συμμορφούνται η πρόταση είτε με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καταγραφεί η πρόταση και οι διοργανωτές συλλέξουν το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Γίνεται μια δεύτερη φάση ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα για την πρωτοβουλία και το τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ενδεχομένω να προκαλέσει προβλήματα. Θα το δούμε παρακάτω. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα τα οποία και εντοπίσαμε. Πρώτον, κάποια οριζόντια θέματα τα οποία παρουσιάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και κάποια άλλα θέματα τα οποία εμφανίζονται αναφάσεις, τα οριζόντια προβλήματα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ε, διάταξη του κανονισμού, ότι οι διοργανωτές θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα που θα οργανώσουν μια επιτροπή, θα συσταθούν σε επιτροπή. τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη, που φέρουν την ευθύνη, όχι μόνο για το πώς λειτουργεί η διαδικασία βάσει του άρθρου 13. Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην οργάνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο, για οποιαδήποτε ζημιά. Αυτό είναι πολύ ευρύος ορισμός και αυτό το παίρνει προσωπικά ο κόσμος αν θα ήταν δυνατόν στην Επιτροπή αυτή να γίνει μια οργάνωση με άλλον τρόπο προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν και νομικά πρόσωπα, θα μπορούσε να αναλυφθεί αυτή η ευθύνη από μια άλλη οντότητα. Αντίστοιχα, τα πρόσωπα, οι διοργανωτές, είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κανόνα προστασίας δεδομένων βάσει του κανονισμού της τρέχουσας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θεωρούνται ελεκτές προσωπικών δεδομένων. Οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει για προσωπικά δεδομένα τα οποία ενδεχομένω να διαρρεύσουν για οποιοδήποτε λόγο είναι στην αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθεί τραπεζικός λογαριασμός, γιατί πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τη χρηματοδότηση του συστήματος της πρωτοβουλίας και για την υποστήριξη που λαμβάνουν. Για να υπάρχει λοιπόν αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να ανοίξει λογαριασμός τραπεζικός στο όνομά τους. Στην παρούσα φάση κάποιες πρωτοβουλίες προσπάθησαν να διοργανωθούν καλύτερα, αλλά στις πιο πολλές περιπτώσεις γίνεται άνοιγμα λογαριασμού σε προσωπικό όνομα και οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει επιβαρύνει τα χρηματικά μέσα του προσώπου αυτού. Όταν συλλέγονται οι πληροφορίες, πάλι παρουσιάζονται κάποια προβλήματα. Άτομα τα οποία δεν είναι παρκώς ενημερωμένα για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Όταν συλλέγουν λοιπόν τις πληροφορίες, το πρόβλημα είναι ότι καταρχάς πρέπει να εξηγήσουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και μετά να ζητήσουν από τους πολίτες να υπογράψουν. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη γνώσης και πληροφόρησης για την πρωτοβουλία. Η υποχρέωση των διοργανωτών να παρέχουν πληροφορίες για την χρηματοδότηση και την υποστήριξη που λαμβάνουν. Δεν εφαρμόζονται σωστά. Και παρά το γεγονός ότι απαιτείται διαφάνεια, η εφαρμογή της διαφάνειας αυτής δεν γίνεται μέσω μιας διαδικασίας όπου η διαφάνεια εποπτεύεται πραγματικά και ελέγχεται. Και αυτό εξαρτάται καθαρά από τις ε, οποιαδήποτε ενστάσεις έχει ο καθής για την έλλειψη διαφάνειας. Αυτά είναι τα οριζόντια προβλήματα που εντοπίστηκαν. Τώρα, για την καταχώρηση της ε, πρωτοβουλίας. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη Γνώσει και πληροφόρηση για την νομική βάση. Πιο πολλοί τρικανοτές αναπτύσσουν προτάσεις και πρωτοβουλίε χωρίς να λαμβάνουν πραγματικά υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει νομοθετικό, νομοθετική βάση. Έχουν την εντύπωση ότι αυτό σχετίζεται με την νομοθεσία και με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν έχει καταρτιστεί ως νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη να βρουν ένα άρθρο στη συνθήκη το οποίο θα αποτελέσει τη βάση του αιτήματό τους, της πρωτοβουλίας τους. Είναι επίσης σαφές για αυτούς ότι για το πεδίο εφαρμογής είναι μόνο νομοθετική πράξη ή για να θίξουν ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Κάτι σαν και αυτό που είπε ο κύριος Τίμερμαντς. Αν ένα θέμα απασχολεί τους πολίτες, ας το συζητήσουμε ακόμα και αν είναι σε πολιτικό επίπεδο και όχι σε νομοθετικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ή σε κάποιο άλλο μέρος. Αυτή η ασάφεια επικρατεί γενικά στο κεφάλι των διοργανωτών. Επίσης, η δυνατότητα που έχουν ε, οι διοργανωτές για να προβούν σε μεταφράσεις, γιατί θα πρέπει τουλάχιστον σε 7 χώρες ε, να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Και η μετάφραση θα πρέπει να είναι σε όλες τις γλώσσες αυτές των 7 χωρών. Αυτό συχνά παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες οι απαντήσεις τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την καταχώρηση δεν είναι εναρμονισμένες. Οι διοργανωτές θεωρούν ότι δεν υπάρχει συντονισμός τόσο μεταξύ της ε, ανταπόκρισης στην πρώτη φάση, που είναι στη φάση της καταχώρησης, και της μετέπειτα απάντησης. Ότι δηλαδή η ανταπόκριση όταν έχουν συλλεχθεί το 1 εκατομμύριο υπογραφές θα μπορούσε να χορηγηθεί εξ αρχή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήξερε ήδη εξ αρχή περί τίνο και το τι αρμοδιότητε έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι δράσεις έχει ήδη λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ένα τμήμα τη πληροφόρηση θα μπορούσε να χορηγηθεί εξ αρχή στου διοργανωτέ. Και ενδεχομένω τότε να είχαν εξετάσει την όλη διαδικασία με άλλο μάτι, να είχαν λάβει άλλες αποφάσεις, να μην είχαν συλλέξει τις υπογραφές. Η επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν στα δύο αυτά βήματα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να συντονιστεί καλύτερα κατά τη συλλογή των υπογραφών. Προκειμένου να συλλεχθούν ε, στο διαδίκτυο, online ε, υπογραφές, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ηλεκτρονικής επαλήθευσης και ηλεκτρονικής υπογραφής. Και έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι δικό της τέτοιο σύστημα. Υπάρχουν δυσκολίες όμως, ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το σύστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα που βλέπετε εδώ. Η συλλογή υπογραφών στα διάφορα κράτη-μέλη αντιμετωπίζει δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, ότι οι απαιτήσει ανά κράτος μέλος διαφέρουν. Χρειάζεται σε κάποιες χώρες ταυτότητα. Από όσου υπογράφουν. Ωστόσο είναι πολύ δύσκολο ένας πολίτης να δώσει τις πληροφορίες του, γιατί ο αριθμός τη ταυτότητα του καθενός θεωρείται ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο που υπόκειται κατά χρήσης. Ο πολίτης δεν έχει έλεγχο. Στο... Δεν μπορεί να ελέγξει πώς θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός δελτίου ταυτότητάς του. Και άρα στις χώρες ε, όπου υπάρχει αυτή η προαπέτηση είναι πιο λίγες πιθανότητες να υπογράψει ένας πολίτης. Δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Άρα η έλλειψη εναρμόνισης αποτελεί πρόβλημα. Όπως και υπάρχουν ε, διαφορές στην ε, έννοια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη Βουλγαρία για παράδειγμα. Κάποιους από τους διοργανωτές, κάποιοι από τους διοργανωτές έπρεπε να καταρτιστούν, να καταχωρήσουν ως ε, ελεγκτές στοιχείων τα άτομα αυτά που βγαίνουν στον δρόμο και προσπαθούσαν να μαζέψουν υπογραφές. Αυτό πήρε πολύ χρόνο και γι' αυτό είχαν πολύ πιο λίγο χρόνο στη διάθεσή τους να συλλέξουν υπογραφές. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται πιο πολύ εναρμόνιση. Σε ό,τι αφορά την επαλήθευση των ε, υπογραφών ε, δεν ε, εντοπίστηκαν πρόβλημα. προβλήματα. Αφού έχει υποβληθεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, το πρόβλημα για τους οργανωτές είναι να αναζητήσει τον λόγο της ακρόασης, την αιτία της ακρόασης, ποιος είναι ο στόχος της ακρόασης. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να, να συζητηθούν και με τα μέλη του Κοινοβουλίου, γιατί τα μέλη του Κοινοβουλίου πιέζουν ε, προωθώντας ανταλλαγές απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν μπορούν σαν παράδειγμα να φέρουν και να χρησιμοποιήσουν εμπειρογνώμονες που θα δώσουν περισσότερες τεχνικές πρωτοβουλίες ή μπορούν να παρέμβουν μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν απαιτείται να υπάρξει μια κάποια διευκρίνηση. Υπάρχουν επιχειρήματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει έλλειψη γνώσεων και είναι πάρα πολύ πιθανό να μην γνώριζαν ότι αν δεν ήταν η πρόταση επιτυχής μπορούσαν να ξεκινήσουν με μία αναφορά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ή θα μπορούσαν επίσης να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρότασή τους και να ξεκινήσει μία νομοθετική πρωτοβουλία με το άρθρο 225 της Συνθήκης. Για αυτά τα προβλήματα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε σε επίπεδο πρακτικό ότι είναι το καλύτερο, είναι να δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία πολιτών, ένα εγχειρίδιο αν θέλετε, που θα περιλαμβάνει και τις απόψεις του Κοινοβουλίου και τις απόψεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έτσι ώστε να δοθεί η απαιτούμενη νομική βοήθεια στους τομείς ε, που είναι προφανώς, ε, προφανές ότι θα απαιτηθεί. Ε, μπορεί να δημιουργηθεί σαν παράδειγμα μια νομική μονάδα η οποία να αναλάβει το ρόλο της ενημέρωσης. Μπορεί αυτή η ομάδα να είναι η μονάδα συγγνώμη να είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, μια μικιό μπορεί να είναι κάτι το επαγγελματικότερο, μπορεί να είναι απλά η εκπροσώπηση των οργανωτών. Συνεπώς λοιπόν ο κανονισμός θα μπορούσε να αλλάξει και τα άρθρα 2 και 3 θα μπορούσαν να διευκρινίσουν καλύτερα το ότι είναι η λέξη οργανωτής, organizer. Τώρα για την καλύτερη τεκμηρίωση των απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης κάποιων από τα άρθρα το άρθρο 4 πιο συγκεκριμένα του κανονισμού. έτσι ώστε να δούμε ε, καλύτερα ποια είναι τα επιχειρήματα και ποιος είναι ο ρόλος του κάθε εμπλεκομένου σε κάθε φάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί τώρα είναι μια, ένα ενδιάμεσο λεγόμενο σύνολο μέσων το οποίο μπορεί να μονιμοποιηθεί αν χρειαστεί και χρησιμοποιείται και κάποιο software αντίστοιχο αλλά αυτό όμως το software θα πρέπει να βελτιωθεί και θα ήταν καλή η λύση το να αναλάβει την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι εμπλεκόμενοι δεν χρησιμοποιούν το μέσο αυτό όσο χρειάζεται και δεν γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας του. Τώρα, ε, οι μεταφράσεις της πρωτοβουλίας η δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν είναι η διαδικασία περίπλοκη η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, Οικονομικής και Κοινομικής Επιτροπής μπορεί να γίνει δεκτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τη διαφάνεια της χρηματοδοτικής στήριξης και στα πλαίσια του Μητρώου Διαφάνειας, αλλά δεν θα πρέπει να μείνει μόνο στα, στις αναφορές παραπώνων. οι οποίες κυρίως έχουν σαν στόχο να σημειώνουν την έλλειψη διαφάνειας και το ότι κάποιες από τις πρωτοβουλίες είναι πολιτικοποιημένες και στηρίζονται κυρίως από πολιτικές ομάδες ή ομάδες εν πάση περιπτώσει οι οποίες έχουν καθαρά πολιτικούς στόχους και δεν είναι ξεκάθαρα διαφανείς. Κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες και κάποιες από αυτές τις συστάσεις όπως είπα θα απαιτήσουν αλλαγές στον κανονισμό, στο άρθρο 11 σαν παράδειγμα, σχετικά με τον στόχο της ακρόασης όπως είπαμε και σχετικά με τους κανονισμούς που θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το άρθρο 11 θα μπορούσε συνεπώς να τροποποιηθεί έτσι ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο γύρω από τον στόχο της πρωτοβουλίας είναι απλά για να προκαλέσει μια νομοθετική πράξη ή να θέσει σε συζήτηση θέματα τα οποία απασχολούν και ανησυχούν τους πολίτες και θα ήθελε ο κόσμος τα ευρωπαϊκά όργανα να τα συζητήσει. Και αυτό μπορεί λοιπόν να αντιμετωπιστεί από τον κανονισμό ως έχει, αλλά μιας και αναφέρεται στη συνθήκη ότι απαιτείται να βρεθεί ε, η μέγιστη δυνατή ε, νομική ε, ασφάλεια. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Α, τον εκπρόσωπο του University College. Είναι δύσκολο, λέει ε, ο κ. Κόεν, να... να παίρνει τελευταίο το λόγο. Ακούσαμε για πάρα πολλές συχνές αλλαγές σε επίπεδο θεσμικό, συνταγματικό κτλ εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά στα πλαίσια της καθημερινότητας του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, στα πλαίσια της νομοθετικής του λειτουργίας και να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά έχουν ανάγκη και από χρόνο και από τεχνογνωσία έτσι ώστε να προωθούν και να εξελίσσουν τα προγραμματά τους. Μα ζητήθηκε λοιπόν να αναφερθούμε στο θέμα της αντιπροσωπευτικότητας των συμφερόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, όλοι οι άλλοι οι οποίοι παρουσίασαν τα προγράμματα τους τα έχουν ολοκληρώσει. Εμείς τώρα το ξεκινάμε. Από τη μία βλέπουμε την προσφορά, το πώς δηλαδή έρχονται οι ενδιαφερόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς κατανέμονται τα ευρωπαϊκά ε, συμφέροντα ε, όπως εκπροσωπούνται βάση περιπτώσει στα πλαίσια του Μητρώου Διαφανείας, στα πλαίσια της οργανώσεως των ακροάσεων και στα πλαίσια των συνεντεύξεων των ενδιαφερομένων. Επίσης ε, θα αναφερθούμε και στον ρόλο των θεσμικών οργάνων και την αλληλοεπίδραση των οργάνων με τα συγκεκριμένα αυτά σύνολα ομάδων συμφερόντων εξετάζοντας επίσης και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την αλλαγή της πολιτικής, όπως επίσης και των συνόλων συνεργασίας, των ομαδοποιήσεών τους, τη συμμετοχή τους σε θέματα όπως οι τριμερείς διάλογοι και το πώς επίσης μπορούμε να εντοπίσουμε αυτά τα συμφέροντα Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα το ποιος εμπλέκεται στη συζήτηση γύρω από ένα πολιτικό θέμα και επίσης ε, να εξετάσουμε ε, είτε το διπλό καπέλο που έχουν μερικές φορές ε, οι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων συμφερόντων σε διάφορες επιτροπές και με διαφορετικούς τίτλους και η συχνότητα επίσης με τις οποίες παρεμβαίνω στους διάφορους τομείς. Αυτά όλα είναι ενδιαφέροντα για τους ε, ευρωβουλευτές να ξέρουν ποιος ασκεί λόμπι, πού ασκεί λόμπι, πώς διαχειρίζεται τη δραστηριότητα αυτή, πώς μπορεί να διευκολυνθεί η επικοινωνία και να διαφοροποιηθεί η συλλογή ε, ε, εκφράσεως απόψεων από διαφορετικά συμφέροντα για να γίνει πιο αντιπροσωπευτική η ενημέρωση και σε ποιο βαθμό μπορεί να προσαρμοστεί το Μητρό Διαφάνειας για να ανταλάβει όλα αυτά υπόψη. Αυτά είναι σε πρόορη φάση. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να υπογραμμίσω είναι ότι κάνουμε μια μεγάλη έρευνα σε όλους τους ε, ευρωβουλευτές και να υπενθυμίσετε κύριε Πρόεδρε ε, και στους ευρωβουλευτές που δεν είναι εδώ το τι ζητάμε να μας πούνε σε ποιους ομιλούν, πώς τους ομιλούν, για ποιο λόγο ε, και να κατανοήσουμε έτσι το τι χρειάζονται οι ευρωβουλευτές για να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια πολιτική άποψη. Και ε, φυσικά κάθε φορά πώς κάνουν αυτή την επικοινωνία σαν εκπρόσωποι μιας επιτροπής, ενός κόμματος, σαν εισηγητές μιας έκθεσης κτλ. Από όλα αυτά θα εξαρτηθεί ο τρόπος με τον οποίο ε, νομοθετούν τελικά. Ε, σε λίγο καιρό, ε, σε ένα χρόνο, θα έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο τα εκφραζόμενα συμφέροντα θα έπρεπε να κάνουν και το τι κάνουν στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπα, σήμερα υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία από την ε, ε, από το Μητρό Διαφάνειας, από, το, από τις στατιστικές, ε, στατιστικές πιστοποίησης. Εδώ θα μπορούσαμε ίσως με κάποιες περισσότερες ερωτήσεις λεπτομέρειες να έχουμε μια πρώτη ιδέα. Βλέπουμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται ακριβώς τα σύνολα έκφρασης συμφερόντων στις Βρυξέλλες Υπήρξαν 6.000 και ε, τέτοιες ομάδες ήδη εγγεγραμμένες, οι οποίες ε, δίδουν στοιχεία στην τράπεζα δεδομένων. Ε, σήμερα άκουσα ότι αυξάνεται ο αριθμός αυτός, έχει φτάσει στο 6.800. Αυτό δείχνει ότι πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι εταίροι είναι δραστήριοι πλέον στις Βρυξέλλες. Οι 6.500 λοιπόν ή 800 ε, με πέντε άτομα, με πέντε άτομα για την κάθε μία από αυτές ε, σημαίνει ότι θα υπάρχουν 30.000 μεμονωμένοι λόμπιστοι οι οποίοι εργάζονται στις Βρυξέλλες. Αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στις Βρυξέλλες ε, σε τομείς όπως το Κοινοβούλιο σε έναν υπάλληλο για δύο λόμπιστ. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς λοιπόν και τις δύσκολες αυτές αριθμητικές συστοιχήσεις θα δείτε από τη μία τις, τα οικονομικά συμφέροντα, τις επιχειρήσεις, τα συνδικάτα, περίπου το 50% των ε, οικονομικών συμφερόντων. Μετά ε, δεύτερο μεγαλύτερο σύνολο είναι η ΜΚΟ και στο τέλος ακολουθούν οι εταιρείε συμβούλων. Ε, Δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί αυτό για να σας δείξω με το pointer πώς λειτουργεί. Ε, φαίνεται ότι εξαρτάται από τη γωνία, αλλά τέλος πάντων δεν τα καταφέρνω. Δεν πειράζει, θα σας τα πω. Ανάλογα με την πολιτική ομάδα, την ομάδα, εδώ αυτά είναι αναπολιτική ομάδα. Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Συνταγματικών Υποθέσεων, όπως κατεβάζουμε έχουμε ε, καταναλωτών, περιβάλλον. Ε, πρόκειται για πράγματα τα οποία εξορισμού έχουν πολύ υψηλή ε, νομοθέτηση, υπάρχει ενδιαφέρον εσωτερικός και 60 με 70% το ενδιαφέροντος που είναι καταχωρημένο για αυτές τις ε, συζητήσεις ε, είναι οικονομική. Ενώ αν δούμε τους καταναλωτές, ε, εκεί είμαστε στο 13%. Επομένως, ανάλογα με τον τομέα, σίγουρα υπάρχει διαφορετικό ενδιαφέρον και επικοινομορφία και είπαμε ότι κάπως αυτά θα πρέπει να τα δούμε όταν συζητούμε τα θέματα αυτά, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα οικονομικά συμφέροντα, θα αλλάξουν τα πράγματα αυτά αν δούμε τις εξωτερικές υποθέσεις, ε, δικαιοσύνη και εξωτερικές υποθέσεις, εκεί αρχίζει να είναι πιο αξιόπιστο το ποσοστό των μη κυβερνητικών οργανώσεων και το τι μπορούν να συνεισφέρουν στη συζήτηση. Και δεν έχω και πολλά πράγματα να σας πω εδώ, αλλά θέλουμε να αναλύσουμε λίγο και τα αποτελέσματα, εξετάσουμε τον τύπο της πολιτικής, αν είναι ε, εκθέσεις ίδιες στο του Κοινοβουλίου και φυσικά βλέπουμε και το φυσικό νομοθετικό αποτέλεσμα της κάθε Γενικής Διεύθυνσης και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει άμεση σχέση ε, και με τις διάφορε, τα διάφορα ενδιαφέροντα, τις δραστηριότητες καθώς επίσης και τις μεγάλες ομάδες ε, εσωτερικώς που συμμετέχουν στους τομείς αυτούς. Υπάρχει μια ενδιάμεση έκθεση την οποία σας δημοσιεύσαμε προσφάτως και αν ενδιαφέρονται κανείς υπάρχουν πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία. Ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το πόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός ε, και πώς αυξάνεται στη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι το Κοινοβούλιο ήταν μια άλλη φωνή, μια διαφορετική εκπροσώπηση συμφερόντων. Εδώ βλέπουμε ότι κάθε δεύτερη μπάρα έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάθε πρώτη μπάρα έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογα με τον τομέα πολιτικής. Έχουμε ε, γεωργία, γεωργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προπολογισμό, προπολογισμό του Κοινοβουλίου κλπ. Ε, και ούτω καθεξής μέχρι κάτω. Και αυτό που δεν μα ενδιαφέρει, όχι σε συνολικά ποσά, αλλά σε ποσοστέ μονάδε, κάθε τομέα πολιτική είναι παρόμοιο. Η μόνη απόκληση είναι ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες εσωτερικές οικονομικές ομάδες στο Κοινοβούλιο και αυτό φυσικά έχει πολύ ψηλότερα ποσοστά ε, εσωτερικά από ό,τι εξωτερικά, αλλά αν το δείτε, τα, οι ομάδες των συμφερόντων είναι παρόμοιες και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει μια αξιόπιστη φωνή, είναι ε, πλέον ο βασικός τόπος ε, ε, προορισμού. Όταν ξεκίνησα εγώ να σπουδάζω, το 30% της πολιτικής διαστηριότητας πήγαινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μικρότερο ποσοστό πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα είναι 50-50 τα ε, στις, ε, από τις ομάδες συμφερόντων. Επίσης, ο τριμερής διάλογος, το γεγονός ότι η πολιτική γίνεται τόσο γρήγορα, αυτό δημιουργεί ενδιαφέρουσες πολιτικές και ενδιαφέροντα δίκτυα. Δεν έχουν εξεταστεί καταλήλως, αλλά ε, ελπίζω να αρχίσουμε να το αντιλαμβανόμαστε στην έκθεση αυτή ε, και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε ίσως να προωθήσουμε. Ε, βλέπω και το ρολόι τώρα και θα προχωρήσω αρκετά γρήγορα. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον και λυπάμαι που δεν μπορώ να σας δείξω εδώ με το δίκτυ. Εδώ έχουμε τις διάφορες ομάδες που έχουμε σε εσωτερικό επίπεδο και σε κάθε επιτροπή για να δούμε ποια είναι η πιθανότητα αν ενδιαφέρεστε για την Επιτροπή Α να συμμετέχετε και στην Επιτροπή Β και Γ και Δ. Αυτό που θέλαμε να δούμε είναι αν οι ομάδες συμφερόντων έχουν τρόπον την περισσότερες πληροφορίες από τους ευρωβουλευτές. Κινούνται σε διάφορες επιτροπές και τι πληροφορίες συλλέγουν αυτοί συνολικά όπως συμμετέχουν σε μια ομάδα. Και πού υπάρχει αλληλοεπικάλυψη συμφερόντων για αυτές τις ομάδες. Δουλεύει. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Ελπίζω ότι θα το δείτε. Αν δείτε πάνω αριστερά, θα δείτε ότι έχουμε πολιτισμό, δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις, εξωτερικέ υποθέσει. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα και είναι πάρα πολύ στενά συνδεδομένα, είναι κοντά στο μηδέν και είναι κοντά στη μηδενική γραμμή. Όσο πιο κοντά είμαστε στο μηδέν, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να συμμετέχετε στην ίδια επιτροπή. Έχουμε λοιπόν εσωτερικές υποθέσεις, εξωτερικές υποθέσεις και πολιτισμό. Σε μια άλλη ομάδα είναι συνήθως η ομάδα που λογικά πηγαίνει στα θέματα οικονομικά, αγοράς ε, και οικονομικής ολοκλήρωσης και μετά έχουμε περιβάλλον και βιομηχανία κάτω αριστερά. Επομένως βλέπετε ότι έχουμε δύο πάρα πολύ ισχυρέ ομάδες και δεν σας εκπλήσει και το γεγονός ότι υπάρχουν και κοινέ αρμοδιότητες, αλληλεπικαλύψεις κλπ. Ε, και αυτό είναι ενδιαφέρον για μας γιατί προσπαθούμε λίγο να δούμε και να διαχειριστούμε τις ομάδες συμφερόντων διότι ορισμένες φορές έχουν ε, πολύ καλύτερες πληροφορίες ε, σε κάποιες γενικές διευθύνσεις ή σε κάποιες επιτροπές από ότι ένας ευρωβουλευτής ή ένας υπάλληλο που προσπαθεί να διαχειριστεί αυτά τα συμφέροντα και πώς μπορούμε να έχουμε και την σχέση μεταξύ των επιτροπών. Εξετάζουμε και τις διάφορες δομές, τις εξωτερικές, κάποιες μη κυβερνητικέ ομάδες έχουν λιγότερους πόρους ή έχουν απλώς ενδιαφέρον για μία μόνο επιτροπή. Έχουμε διάφορες ομάδες, ε, μία μικρότερη είναι ανάμεσα στην ανάπτυξη και στο εμπόριο, αλλά εκεί οι δεσμοί είναι λίγο ε, πιο αποδυναμωμένοι. Αυτή τη διαφάνεια θα την αφήσω. Στους ανεπίσημους λοιπόν κανόνες έχουμε πιο πολύ δυνατότητα πρόβλεψης ε, σε ακροάσεις, όχι συνεμερινές συνεδρίσεις. Ε, και αυτό παίρνει πολύ χρόνο και ο Άλεξ, ε, ο υπεύθυνο για την έρευνα, χρειάστηκε να πάει. Είχαμε 2.080 ομιλητέ που έχουν προσκληθεί σε 281 εκδηλώσει σε πολλά κοινοβούλια. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο και πιο πολλές ακροάσεις ε, να γίνονται και πιο, μη, πιο πολλούς μη θεσμικούς ομιλητές που προσκαλούνται. Αυτό μπορείτε να θεωρήσετε ότι αποτελεί την απόρρια της επιθυμίας να ακούσουμε με εναλλακτικέ φωνές. Πιο πολλούς ακαδημαϊκούς, πιο πολλά think tanks. Η Λίμπε κάλεσε τους ε, πιο πολλούς μη θεσμικούς φορείς, πάνω από 350. Και είχε 900 άτομα προσκεκλημένα στην Επιτροπή. Κάτι άλλο που κάνουμε για τη συλλογή δεδομένων. Κοιτάμε ε, εκθέσεις και εισηγητές 5 επιτροπών για 7 κοινοβούλια, 300 ε, εκθέσεις εξετάσαμε. Λιγότερο από το 2% έχουν καταγράψει Εμπλεκόμενε φορείς. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι η πρώτη λοιπόν ε, σύσταση, πολύ εύκολη. Ο αριθμός εμπλεκόμενων φορέων που αναφέρονται θα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό είναι το γράφημα όσων εμφανίζονται πιο συχνά που αποτελούν συχνούς συνομιλητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμπορικά συνδικάτα, ενώσεις καταναλωτών. Άρα αυτοί είναι οι παραδοσιακοί συνομιλητές. Ποιοι είναι όμως οι λιγότερο συνηθισμένοι που θα περίμενε κανείς ότι έρχονται στο, κοινοβούλιο. Να κλείσω λέγοντας ότι συνολικά το, το μήνυμα είναι πολύ θετικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ε, κάποιος ε, μελετήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη ΣΥΠΑ και τι γίνεται με τις ομάδες πίεσης, είστε πάρα πολύ διαφανείς σε σύγκριση με αυτά. Ε, είναι κάποιες ομάδες άσκησης πίεσης που εξακολουθούν να αυξάνονται. 300 τα 300 τέτοιες ομάδες έχουν προσταθεί προσφάτως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το... η πλατφόρμα για την άσκηση πιέσεων μετά τη Λισαβόνα. Αυτό είναι καλό. Βλέπουμε λοιπόν μια οριμότητα, μια πιο επαγγελματική διαμόρφωση των συμφερόντων, μεγαλύτερη διάδραση μεταξύ των ομάδων και των βουλευτών. Αν αυτό όμως το αποδεχτούμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτή της διαφάνειας, ε, διαφοροποίησης αυτής και πώς μπορεί να βελτιωθεί η διαφοροποίηση και η πρόσβαση. Κάποιες προσωρινές συστάσεις, προσωρινές μόνο το τονίζω. Καταρχάς, κάτι που έχω ακούσει στη συζήτηση του τελευταίους μήνες, ότι το, ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διευκολύνει κάποιες ομάδες και να βοηθήσει να χρηματοδοτήσει κάποιες ομάδες να συμμετάσχουν για να βελτιωθούν οι δραστηριότητε μεταξύ των επιτροπών. Αυτό προέκυψε από τις δραστηριότητε που εξετάσαμε. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία και συντονισμός σε ό,τι αφορά την διαφάνεια και την νομιμότητα. Θα μπορέσετε να λάβετε πληροφορίες για διαπιστευμένες και μη ομάδες πίεση και να τι δημοσιεύσετε. Μιλούσα πριν από πολλά χρόνια για το Diane Wallins για να εκτήρουν μητρό οι βουλευτέ. Αυτό αποτελεί μια λύση, μια ιδέα. Όχι λεπτομέρειε, αλλά το άτομο το οποίο ήρθε και του επισκέφτηκε. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε επίση να εξετάσει αύξηση διαφάνεια διαφάνειας τα δεδομένα αυτά. Η βάση δεδομένων είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη διαχειριστεί κανείς. Την καθαρίσαμε επί μήνες. Ίσως κάποιος θα μπορούσε να βελτιώσει την διαπαφή για να μπορεί να είναι προσβάσιμη στο κοινό. Το νομοθετικό αποτύπωμα. Ξέρω ότι συζητιέται εδώ και πολύ καιρό, πολλά πολλά χρόνια εδώ στις Βρυξέλλες αυτό. Και αυτό μπορεί να ταιριάξει και με την συζήτηση που είχαμε με τον Αντιπρόεδρο Τίμπερμαντ προηγουμένω. Μπορούμε να ζητήσουμε κατά πόσον θέλουν να συμμετάσχουν. Όχι μόνο να δηλώνουν κατά πόσον είναι διαπιστευμένοι, αλλά να λένε ότι πηγαίνω στην ΧΥΠΣΗ επιτροπή, στη ΧΥΠΣΗ γενική γραμματεία, στη ΧΥΠΣΗ γενική ε, μόνιμη προσωπία. Να καταγράφουν δηλαδή όλες τις επαφές που κάνουν. Και θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε να δηλώνουν κατά πόσο έχουν διπλή ιδιότητα. Ως εμπορική ένωση, ως εκπρόσωποι ε, εταιρεία, ως μέλη think tanks μπορεί να έρχονται να μας μιλήσουν, να αναφέρουν όλα τους τα συμφέροντα, όλα τα φόρουμ τα οποία εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή. Ανανέωση των δεδομένων. Είπαμε ότι έχουμε 300 νέες οργανώσεις τους τελευταίους μήνες μόνο. Αλλά κάποιοι από τους παλιούς δεν έχουν ανέωσει, δεν έχουν ενημερώσει τα στοιχεία τους από τη στιγμή που καταχωρίστηκαν. Θα πρέπει λοιπόν τα στοιχεία τα οικονομικά να ενημερωθούν. Μπορεί να είναι ίδια, όπως και παλιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ενημερώνονται. Και τέλος, μπορούμε να ασκήσουμε επίσης στους βουλευτές και στους υπαλλήλους να επικοινωνούν με πιο ευνοϊκό τρόπο με όσους είναι καταχωρισμένοι, γιατί στην παρούσα φάση δεν γίνεται αυτή η διάκριση. Ίσως λοιπόν να μπορούσε κανείς να έχει ένα πρώτο δικαίωμα προνομιακό επαφής σε περίπτωση που κάποιος είναι καταχωρισμένος. Δεν το έχω σκεφτεί καλά αυτό ακόμα, αλλά θα μπορούσαμε να βρούμε κίνητρα για να καταχωριστεί ο κόσμος και για να απαντήσω το ερώτημα για το κατά πόσο θα πρέπει και το Συμβούλιο να μπει στην βάση δεδομένων. Είναι δύσκολο αυτό γιατί, όπως ξέρουμε, κάνει πολύ, γίνεται πολύ lobbying στο Συμβούλιο, ασκείται πολύ πίεση. Αλλά ακόμα και αν ε, συμμετείχε στο Μητρό Διαφάνεια, το πρόβλημα είναι, θεωρώ, πώς θα πιάναμε το εθνικό λόμπι και αυτό που ανακύπτει από αυτό στον Ηνωμένο Βασίλειο, το Μητρό Συμφερόντων και στη Γερμανία νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα. θα υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές λοιπόν σε αυτά που θα ξέραμε ένα χώρα για το εθνικό λόμπινγκ. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει η πρόοδος. Ε, δεν ξέρω αν η κυρία Κάουφμαν ε, θέλει να θέσει μια ερώτηση, ίσως να υπάρχει κάποιοι που... Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε, ναι. Όχι, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για το θέμα του ECI, αν μου επιτρέπετε. Και θα μιλήσω γερμανικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρόβλημα με την σημερινή μας αχρόαση, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά και διαφορετικά θέματα τα οποία και επεξεργαζόμαστε από εκείνου και για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είχα προετοιμαστεί γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Επειδή έχει περάσει και η ώρα θα περιοριστώ σε κάποιες περιορισμένες παρατηρήσεις. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς και στην ακρόαση και σήμερα. Ότι καλό θα ήταν και σημαντικό θα ήταν να είμαστε λίγο λιγότερο τυπολάτρε σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Να αναζητήσουμε πιο πολύ τον πολιτικό διάλογο. Αυτό με απασχολεί πάρα πολύ, ξέρετε, γιατί έχουμε πάρα πολλέ περιπτώσει. Έχουμε μάλλον διάφορε περιπτώσει όπου θα θέλαμε να λάβει σοβαρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συμφέροντα που εκφράζονται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, μια πρωτοβουλία η οποία πέτυχε τα δικαιώματα των μειονοτήτων και είχε ευρεία υποστήριξη. Το TTIP, ένα πολύ γνωστό θέμα, το οποίο υποστηρίζουν 320 μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Κατά δεύτερον, να συμφωνήσω με την ε, ερώτηση που έθεσε η συνάδελφος Ρέντινγκ. Πολύ δικαιολογημένη και θα έπρεπε να το τονίσουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά όσα μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρωτοβουλία των Πολιτών, θα πρέπει να σκεφτούμε την αναθεώρηση του κανονισμού. Υπάρχει ανάλυση την οποία ακούσαμε σήμερα και θα ήθελα εκ βάθους καρδίας να σας ευχαριστήσω για τα πολύ επακριβή και λεπτομερή εργασία που κάνατε και που μας βοηθάει ιδιαίτερως. Η Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων ε, εντατικά παρακολούθησε το θέμα αυτό και θα μας αναφέρει τα σχετικά η διαμεσολαβήτρια. Υπάρχει ένα δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων που παρακολουθεί το θέμα αυτό επισταμένως και όπου διαρκώς γίνονται εργαστηρία και η αλυσίδα των προβλημάτων που ακούσαμε εν μέρη σήμερα είναι πολύ μακριά Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τις λεπτομέρειες. Αν θέλουμε, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει όλους να μας απασχολεί, αν θέλουμε όντως να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και το μέσο, το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών κινείται προς την κατεύθυνση αυτή που θα θέλαμε όλοι, ε, τότε χρειαζόμαστε αλλαγή, επιγόντως αλλαγή στον κανονισμό. Γιατί άλλο μπορεί να μαραζώσει το εργαλείο αυτό. Έχουμε ακούσει τα αριθμητικά στοιχεία και να προσθέσω και το εξή. Μόνο τέσσερι πρωτοβουλίε πολιτών βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα και πάνω από το ίμιση όλων των πρωτοβουλίων που έχουν κρατεθεί έχουν απορριφθεί ή αποσυρθεί. Δεν έχει λειτουργήσει καθόλου. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν επακριβώς και νομίζω ότι αυτό είναι το συμπεράσμα της μελέτης, να δούμε ως ε, Επιτροπή να μιλήσουμε και ως Κοινοβούλιο να συζητήσουμε τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για να δούμε πώς έχει λειτουργήσει η πρωτοβουλία από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός. Δεν επαρκούν τα όσα έχουμε πετύχει. Θα πρέπει λοιπόν το εργαλείο αυτό εκ νέου να το κοιτάξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου, μιας και δεν υπάρχει κανένας άλλος, να κάνω κάποιες ερωτήσεις, να θέσω μία ερώτηση για αυτό που είπατε ότι για να υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα, ότι πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα γιατί αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία. Να ρωτήσω λοιπόν σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή δυναμική των ε, πολιτικών κομμάτων, ομάδων, αλληλεξαρτήσεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πολιτικά κόμματα, το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ε, διαδραματίζει πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο ρόλο για την ε, δημιουργία διεθνικών δημοκρατιών, γιατί αυτή είναι η ευρωπαϊκή παράδοση. Τώρα έχουμε κόμματα που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διαφορετικούς σχηματισμούς. Αυτό συμβάλλει στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η απάντηση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ναι, η απάντηση είναι καταφατική όπως σας είπα. Τα θέματα τα οποία αντιμετώπισε το Κοινοβούλιο πριν από 35 χρόνια δεν είναι τόσο πιεστικά σήμερα, αλλά είναι πιεστικό το θέμα το ότι περιμένουμε πιο πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Η απάντηση είναι ναι, καταφατική, αλλά κατά πόσο επαρκεί αυτό. Και εκεί βρίσκεται το κλειδί. Αυτή είναι η ερώτηση κλειδί, αν θέλετε. Ειλικρινά δεν έχω απάντηση να σας δώσω, γιατί θα χρειαζόμασταν εκτενέστατη μεταρρύθμιση. Δυστυχώ δεν ήμουν εδώ σήμερα το πρωί, δεν είχα αεροπλάνο. Δεν μπορούσα να πάρω πιο νωρί αεροπλάνο, πιο πρωινή πτήση. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτό που εξετάζουμε είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και ναι και όχι, λοιπόν, είναι η απάντηση. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί φυσικά οι εμπειρίες μου διαφέρουν ανά χώρα, αλλά και τότε από στο εθνικό επίπεδο δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η δίωδο επικοινωνία για την Ευρώπη που περνάει από κομματικέ ε, από οδούς Όταν πηγαίνουμε στις πα, παρτίδες μας, πα, πατρίδες μας, δεν ε, πουλάμε σε επίπεδο κόμματο στην Ευρώπη, στον κόσμο. Δεν συμβάλλουμε έτσι στην αύξηση της ευαισθητοποίησης. Εκεί κάτι λείπει, έχω την αίσθηση, στο τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας των οδών αυτών. Δεν σημειώνουμε τα αποτελέσματα που θα μπορούσαμε να σημειώσουμε σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της Ευρώπης στον πολίτη. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Ήταν πραγματικά σταρπαστικά όλα όσα μας είπατε για τις πληροφορίες. Δεν νομίζω ότι στο, στο Κοινοβούλιο αντιλαμβανόμαστε πόσο σε βάθος περνάνε οι ακαδημαϊκές αυτές μελέτες. Θα έπρεπε να κάνουμε πιο πολλές από αυτές τις συζητήσεις. Uh, και δεν ξέρω αν θα ήθελε κανείς να σχολιάσει, γιατί έχω και άλλη μια ερώτηση να κάνω. Αυτό που άκουσα από κάποιον Βρετανό, ότι οι ευρωπαϊκές ε, πολιτικές προχωράνε τόσο γρήγορα, πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Γιατί είναι τόσο διαφορετική εικόνα που έχουμε. Εσείς ε, στο τέλος συγκρίνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, κάτι τέτοιο. Από πού προκύπτει αυτό το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, από πού προέρχονται αυτές οι ομάδες συμφερόντων. Αρχίζουν να απομακρύνονται από το εθνικό επίπεδο γιατί όλο και περισσότερες ε, εθνικές πολιτικές ε, ε, προέρχονται από την Ευρώπη ή είναι μία αλλαγή, έχουμε λιγότερο στο Λονδίνο και περισσότερο στο Βερολίνο, ξέρω εγώ κλπ. 20 χρόνια που μελετάω τα λόμπι στην Ευρώπη ξεκίνησα από την ενιαία αγορά και τότε είχαμε τα εθνικά λόμπι που ερχόντουσαν εδώ και άρχιζαν να μαθαίνουν σιγά σιγά να ε, έρχονται σε επαφή με τις Βρυξέλλες. Αλλά σιγά σιγά έγιναν πιο επαγγελματικά τα πράγματα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ λόμπι, το οποίο είναι μοναδικό για τις Βρυξέλλες. Προσφάτως μιλούσα στη Washington για το θέμα αυτό και δεν μπορούν να αντιληφθούν τη συνένεση. Υπάρχει συνένεση παντού, αλλά δημιουργείται συνεχώ. Είτε είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε στο Κοινοβούλιο. Οι ομάδε πρέπει να βρουν κάποιο κοινό έδαφο να δημιουργήσουν συμμαχίε. Και γιατί αυτό είναι το θέμα της αξιοπιστίας των πληροφοριών που έχει σημασία και η σφαίρα επιρροή των πληροφοριών, ε, η αξιοπιστία σου προκύπτει από αυτό είναι τελείω διαφορετικά. Ε, στη Washington τα πράγματα είναι περισσότερο με βάση το χρήματα ε, και στην Ευρώπη δεν λέω ότι είμαστε αφελεί. Ε, φυσικά και έχουν σημασία τα χρήματα. Αν έχουμε 10 λόμπι και έχει και μία ε, εταιρεία συμβούλων και μια νομική εταιρεία, ε, τότε σίγουρα θα έχουμε και μια τεχνική έκθεση που μπορεί να επηρεάσει ίσως λίγο περισσότερο στην Επιτροπή ή οπουδήποτε αλλού, αλλά οι Βρυξέλλες είναι θέμα αξιοπιστίας ε, και οι υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μένουν οι ίδιοι ε, για πάρα πολλά χρόνια και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται για παράδειγμα με ένα θέμα είναι ίδιοι και ξέρουν πάρα πολύ καλά οι, τα λόμπι σε ποιον μπορούν να μιλήσουν και σε ποιον δεν μπορούν να μιλήσουν. Υπάρχουν και κάποιοι ευρωβουλευτέ που έχουν δημιουργήσει συγκεκριμένη θεσμική μνήμη, τα λόμπι. Πρέπει να προσέξουν λοιπόν πάρα πολύ τη φήμη που έχουν δημιουργήσει, αν θα μπορέσουν να την ε, διατηρήσουν ή να την καταστρέψουν. Είναι λοιπόν ένα μοναδικό φαινόμενο το λόμπι των Βρυξελών, δεν ομοιάζει με αυτό του Λονδίνου και τον, ε, του Βερολίνου ή οποιοδήποτε άλλο, διότι είναι προσαρμοσμένο στις θεσμικές μορφές που έχουμε εδώ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, γιατί έχουμε τόσο πολύ λόμπι, γιατί έχουμε τόσα ε, τόσες πολλές ομάδες, 6.500 ομάδε, ε, καταχωρισμένες ομάδες. Διότι οι περισσότεροι κανονισμοί, η περισσότερη νομοθεσία προκύπτει από τις Βρυξέλλες. Και ε, τέλος πάντων ε, πας εκεί που σε πάει το ρεύμα, εκεί που θα γίνει η πολιτική, εκεί που μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Επίσης μπορεί να ακολουθήσεις και τις ε, τάσεις πολιτικής και να πας σε εθνικό επίπεδο από εκεί και πέρα και να πρέπει να εφαρμόσεις νομοθεσία σε τηλεπικοινωνίας. Αλλά τα πάντα ξεκινούν από, δουν και, από εδώ και επιχειρήσεις το γνωρίζουν και αφιερώνουν πολλούς πόρους και χρόνο για να στελεχώσουν τα ευρωπαϊκά τους γραφεία και να έχουν μια ομάδα που να μπορεί να ανταποκριθεί και να έρθει εδώ στις Βρυξέλλες. Είπατε κι εσείς ότι για το Συμβούλιο είναι μεγάλη πρόκληση, διότι άκουσα και κάποια σχόλια ότι Ακόμα και οι υπουργοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν λομπίστε, άμα έρχονται εδώ να προσπίσουν τα εθνικά του συμφέροντα. Επομένω, είναι μεγάλη πρόκληση για μα. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Κάναμε λάθος, ε, πρέπει να το ομολογήσω που σας βάλαμε όλους εσάς σε μια μέρα. Κανονικά πρέπει να γίνει μια εβδομάδα συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα θέματα και είναι πολύ σημαντικά τα όσα ετοιμάσατε και πραγματικά αν είχαμε και πιο ε, πλήρε εκδοχές των, όσων ετοιμάσατε, δεν ξέρω τι κάνει το τμήμα πολιτικής, αλλά θα χρειαστούμε και την εμπειρογνωμοσύνη σας, διότι τώρα ξεκινούν οι εργασίες μας και πραγματικά... Ε, θα γίνουν σοβαρές εργασίες σε όλα τα διαθεσμικά ζητήματα και αυτά που συζητήσαμε σήμερα το πρωί, ανάλυση των αλλαγών επίσης, ε, ε, θα εξετάσουμε τα θεσμικά όργανα εκ των έσω για την αποτελεσματικότητά τους και είναι πάρα πολλά. Και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας, ίσως αργότερα, και θα σας ε, κάνουμε και θα σας ζητήσουμε αυτά που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας αφήνετε με πληθώρα πληροφοριών και πολύ τροφή για σκέψη. Ε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήρθατε εδώ σήμερα και για την υπομονή σας. Τα πάντα είναι μέσω ε, διαδικτύου. Μην νομίζετε ότι φύγαν όλοι. Ε, τα πάντα μέσω διαδικτύου. Δεν το, θα χρησιμοποιηθεί αυτό εναντίον σας, αλλά ό,τι πείτε θα μείνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρασε τη συνεδρία σας.